Possiamo cominciare i nostri lavori. Preliminarmente informo, come d'abitudine, come normalmente, che la nostra seduta è. Όπως γνωρίζετε συνήθως μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε κάθε φορά η ημερήσια διάταξη έχει διανεμηθεί ήδη από τις 14 του μηνός και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρείται δεκτή. Θα τεθούν ορισμένες ερωτήσεις στο σημείο 11 για την έκθεση Τρασκόφσκι. Αν ε, είναι δυνατόν θα το κάνουμε λοιπόν αύριο το πρωί αυτό. Λοιπόν δεν ακούγεται κάποια αντίρρηση, συνεπώς θεωρείται δεκτή η μερίσια διάταξη. Στο φάκελο θα βρείτε το τελικό κείμενο της ε, υπηρεσίας τεκμηρίωσης σχετικά με την κατάσταση και το στάδιο των διαδικασιών επικύρωσης. Επί τη βάση αυτού του εγγράφου θα δούμε την μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο των ε, Κοινοτικών Συμφωνιών. Σήμερα θα ασχοληθούμε λοιπόν με το θέμα αυτό μέσω της ε, δημόσιας ακρόασης για την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας στο κομμάτι το οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες που ανταποκρίθηκαν στην πρότασή μας και θα εμβαθύνουν στο θέμα αυτό. Ένα θέμα το οποίο βέβαια έχουμε αντιμετωπίσει επανειλημμένα και το οποίο εισηγητής είναι ο συνάδελφος Ράγκελ. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Αντώνιο Βιτορίνο, πρόεδρο της Notre Hope και τέος κοινοτικό επίτροπο εδώ και κάποια χρόνια. Έχουμε τον καθηγητή Ίγκολφ Πέρνιτσε, Πέρνισε, διευθυντού του Ινστιτούτου Βάλτερ Χάλσταϊν του Πανεπιστημίου Χούμπολ του Βερολίνου. Τον έχουμε συναντήσει ήδη ε, σε ένα σεμινάριο στις Βρυξέλλες και στην πόλη του. Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή Νίμαντ Κρίστενσεν που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα είναι παρόν για λόγους ε, ε, ανηλυμένων υποχρεώσεων ο καθηγητής κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης του European Policy Center, του EPC, που έχει πάρει μέρος σε άλλα σεμινάρια βέβαια. Έχουμε όμως ανάμεσά μας τον καθηγητή Στέβεν Μπλόκμαν του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικών Επιστημών και τον καθηγητή Ρόντρικ Πάρξ, ο οποίος είναι μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων της Βαρσοβίας. Ο γραμματέα μου θύμισε να θυμίσω και το όνομα του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο είχα κάνει όμω από πριν. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα τεθεί είναι θα έλεγα η στροφή την οποία έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή που πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερο βάρος στο κοινοβουλευτικό κομμάτι και λιγότερο στο λεγόμενο εκτελεστικό προεδρικό. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον συνάδελφο Ραντζέλ. Uh, να σας καλωσορίσω όλους σήμερα ε, για αυτή την πρώτη συνάντηση. Έχω εδώ δίπλα μου τον κύριο Βιτορίνο, τον οποίο ήδη παρουσιάσατε. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσει κανείς σε αυτή τη φάση σε μια μακρά παρουσίαση της συγκεκριμένης έκθεσης. Γιατί έχει επανειλημμένα συζητηθεί στην Επιτροπή μας. Το περιεχόμενο της εκθέσεως είναι θα έλεγα γνωστό, όπως γνωστές είναι και οι αντιθέσεις τις οποίες προκαλεί. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σας και την προσοχή των ε, εμπειρογνωμόνων που είναι παρόντες Τους βασικούς στόχους θα έλεγα που έχει αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας θυμίζω. Η πρώτη έκθεση, ο πρώτος στόχος μάλλον, είναι να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε, να δημιουργήσουμε αν θέλετε ένα ιδεολογικό σχήμα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται το Κοινοβούλιο στις διάφορες προβλέψεις και άρθρα της συνθήκης. Να μην αγνοούμε εδώ ότι κινούμεθα ακόμα στο πλαίσιο των σχέσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός είναι ο κεντρικός μας προσανατολισμός. Η βασική ιδέα λοιπόν δεν είναι μόνο να προχωρήσουμε σε, μια διάγνωση της κατάστασης την οποία αντιμετωπίζουμε, αλλά να ε, προετοιμαστούμε και για την ε, έναρξη των εργασιών της νέας Επιτροπής μέσω του διορισμού των Επιτρόπων και του Προέδρου της. Βασικός μας στόχος λοιπόν και ξεκάθαρος θα έλεγα στόχος είναι να καθορίσουμε την θεωρία η οποία θα στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο τον μήνα που θα ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εκλογές, μετά το Μάιο δηλαδή. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να αναλύσουμε την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα και θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε ένα κάποιο ιδεολογικό σχήμα θα έλεγα, την ερμηνεία όπως σας είπα και προηγουμένως, την οποία θα δώσει το Κοινοβούλιο στα κείμενα τα οποία προτείνονται κατά τη διάρκεια της περίοδου διαπραγμάτευσης. Είναι περιορισμένη ίσως η εμβέλεια αυτής της προσπάθειας, αλλά θυμίζω ότι για πρώτη φορά η συνθήκη της Λισαβόνας θα εφαρμοστεί στους συγκεκριμένους αυτούς τομείς, δηλαδή του διορισμού της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου το θέμα παρουσιάζεται πολύ σημαντικό. Δεύτερον, θα θέλαμε να ασχοληθούμε και με κάποια προβλήματα τα οποία περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο Επιτροπής Κοινοβουλίου και τα οποία άπτονται φυσικά των διοργανικών σχέσεων. Υπάρχουν και ορισμένες επιπλέον προβλέψεις οι οποίες αφορούν στο Συμβούλιο. Και οι προβλέψεις αυτές ε, ίσως ε, θα πρέπει να μας οδηγήσουν ε, στην αναθεώρηση της διοργανικής που θυμίζω ότι λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια με το ίδιο πλαίσιο ή μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Από το 2003 δηλαδή μέχρι και τώρα σε ένα πλαίσιο νομοθετικής συνεργασίας ή καλύτερα συνεργασίας ε, του νομοθετικού με το εκτελεστικό. Δεύτερο θέμα είναι βέβαια να μείνουμε στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και των διαπραγματεύσεων των συνθήκων και των συμβάσεων με τους ε, τρίτους εταίρους. Ποιος είναι εδώ ο ρόλος του Συμβουλίου και κυρίως του Κοινοβουλίου. Και ένα επιπλέον θέμα είναι ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μία σχέση ε, πραγματικού διαχωρισμού των εξουσιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γαλήνιο θα έλεγα στις σχέσεις μας με τις χώρες μέλη. Δεν είναι καν σαφές το τι επιθυμούμε στην παρούσα φάση αλλά το να ενισχύσει κανείς την νομιμότητα και την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών οργάνων δεν θα σημαίνει σε καμία περίπτωση την αντίστοιχη μείωση κάθε ενός οργάνου. Ε, και γι' αυτό ακριβώς είμαι θα ιδιαιτέρως επιφυλακτική στην προσπάθεια διαμόρφωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή έχει σαν παράδειγμα μεγάλη σημασία να υπάρχει δυνατότητα λογοκρισία σε εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει, των συζητήσεων σε άλλο όργανο μέσω ναι, ειδική πλειοψηφία και όχι μόνο, μόνο ομοφωνίας, όπως επίσης και το... So there is also here a quite clear trend of trying to shape uh, uh, a separation of powers. Ε, εν πάση περιπτώσει και με απλή πλειοψηφία θα μπορεί να τεθεί εν πάση περιπτώσει το θέμα αναδιακοπή διαδικασία από πλευρά του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ο βατικός στόχος λοιπόν να προσπαθήσουμε από τη μία να διαμορφώσουμε μια σταθερή λογική στήριξη των θέσεών μας αμέσως μετά τις εκλογές να επιλύσουμε κάποια θετικά, ε, ε, τεχνικά θέματα όπως ε, το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων, των εφαρμοστικών πράξεων, να αντιμετωπίσουμε το θέμα της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή και τέλος το λεγόμενο ιδεολογικό λίγο αν θέλετε θέμα του διαχωρισμού των εξουσιών με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας όπου υπάρχει σύγχυση των εξουσιών υπάρχει σύγχυση και στον τομέα της δημοκρατίας. Αυτές είναι οι ιδέες μου λοιπόν και γι' αυτό θα ήταν χρήσιμο να ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων και δίνω το λόγο αμέσως στον φίλο Αντώνιο Βιτορίνο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγητά, κύριε και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην πρόκλησή σας, λαμβάνοντα υπόψη ορισμένα από τα βασικά θέματα που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως σε τρία. την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον πολιτικό ρόλο και αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τις σχέσεις των δύο οργάνων σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές εξουσίες. Παρ' αυτά, να μου επιτρέψετε προκατακτικά να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση. Πιστεύω ότι στο προσεχές μέλλον το κύριο χαρακτηριστικό της θεσμικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα είναι κάτι που προ 15 ετών αποκαλούσε ο Ζακ Τελόρ διαφοροποίηση. Η Ευρωζώνη, οι χώρες δηλαδή που είναι στην Οικονομική και Ένωση, Πρόκειται να γίνουν ο πυρήνας μιας σε βάθος οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης. Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση είναι η κύρια πολιτική της Ένωσης, αλλά Δανία και Ενωμένο Βασίλειο με απόκληση στόχων τους επιτράπει από την συνθήκη Μάστριχτ να τους έχουν στόχους αυτούς, αλλά πρακτικά η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα εξελιχθεί και θα βαθύνει ακολουθώντας μια λογική στενή συνεργασία με ένα σύνολο κανόνων και υποχρεώσεων, δεσμεύσεων που θα δεσμεύουν συγκεκριμένη ομάδα χωρών μελών, εκείνων δηλαδή που έχουν το κοινό νόμισμα και που υποχρεούνται και που μπορούν μάλλον να συμμετάσχουν, να ε, ε, ε, χρησιμοποιήσουν και αυτές το ευρώ, το ευρώ, όταν θα, θα πληρώνουν τα κριτήρια. Αυτά μέχρι τώρα έχουν γίνει στη βάση διακυβερνητικών συμφωνιών. Όμως, πιο σημαντικό από την νομική βράση είναι αυτό που διακυβεύεται από την θεσμική άποψη είναι το ερώτημα πώς να διασφαλίσει κανείς την ακαιρεότητα του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης της, Ευρωπα... της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ιδίως δε τα νομοθετικές εξουσίες του Κοινοβουλίου, την εξουσία πρωτοβουλία της Κομισιόν και βέβαια τον δικαστικό έλεγχο που ασκεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το βάθεμα αυτό της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης θα προκαλέσει εντάσεις, ίσως και συγκρούσεις μεταξύ των όσων πρέπει να γίνουν στο επίπεδο των 18 χωρών μελών των 28 χωρών μελών μάλλον και του πυρήνα που είναι οι χώρες που συμμετέχουν μόνο στη ζώνη ευρώ. Γι' αυτό νομίζω ότι η ακαιρεότητα των θεσμών και το να βρεθούν στο επίκεντρο, στο προσκήνιο οι θεσμοί, αυτό θα είναι θεμελιώδους σημασίας για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ενδεχόμενες σύγκρουσεις τώρα. Έχοντας πει αυτά τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι σαφές και ιδίω για το Κοινοβούλιο ότι αποκλείεται απολύτως να δημιουργηθεί οποιοδήποτε παράλληλο θεσμικό πλαίσιο αποκλειστικά για την ζώνη ευρώ. Εκτός δηλαδή του πλαισίου που ήδη υφίσταται. Ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να βαθύνει η νομισματική ένωση θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες προσαρμογές των υφισταμένων θεσμών. Για παράδειγμα, η δυνατότητα δημιουργίας μιας υποεπιτροπής οικονομικών και νομισματικών θεμάτων της, ε, της Επιτροπής ΕΚΟΝ του Ευρωκοινοβουλίου, όπου γνωρίζω ότι εδώ βέβαια δεν σημειώνεται συνένεση μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι μια ειδική δομή εντός του Κοινοβουλίου που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου μέσα από τη δυναμική του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τη δυναμική που έχει ξεκινήσει με το άρθρο 13 του ε, Δημοσιονομικού Συμφώνου θα είναι κέρια για να μπορέσει να αναπτυχθεί η σχέση και μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων των χωρών μελών. Μετά από αυτή την προκατακτική παρατήρηση για την διαφοροποίηση και για τις θεσμικές επιπτώσεις της, να επιστρέψω στην πολιτική νομιμοποίηση της Κομισιόν. Όπως είπε ο εισηγητής Πολ Ραντζέλ, πρέπει να ξεκινήσουμε ένα νέο σύστημα, ένα νέο μοντέλο, και πρόκειται να το κάνουμε αυτό βέβαια, για τον ε, διορισμό του Προέδρου. Το μοντέλο αυτό εγκρίθηκε ήδη από την συνέλευση τότε, και βλέπω πολλά πρόσωπα γνωστά από τότε εδώ, είχαν προταθεί διάφορες εναλλακτικές επιλογές, που είχε απορριφθεί, είχαν απορριφθεί ορισμένες, έτσι δεν υπάρχει καμία διασύνδεση ανάμεσα στην εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν και στα αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια διασύνδεση στο οικείο άρθρο, αλλά το θέμα είναι πώς θα υλοποιηθεί η διασύνδεση, ο σύνδεσμος αυτός, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο θα πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, όταν θα κληθεί να διορίσει τον υποψήφιο για την Προεδρία της... εφόσον αυτός θα έχει εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα βήμα για να υλοποιηθεί ο σύνδεσμος αυτός έχει ήδη ληφθεί από διάφορες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου όταν αυτές ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν υποψηφιότητες για την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τις ευρωεκλογέ. Αυτή η ιδέα βεβαίω είχε διατυπωθεί ήδη προ 15 ετίας από τον τότε Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ. Ο στόχος του συνδέσμου αυτού είναι να δώσει ένα πρόσωπο, να βάλει ένα πρόσωπο σε ένα πολιτικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν οι πολίτε να συμμετάσχουν στις εκλογέ. Ανατρέποντα έτσι την φθήνουσα τάση συμμετοχή στι ευρωεκλογέ. Έλαβαν λοιπόν την απόφαση πλήρωνε πολιτικέ ομάδε και δίνουν έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βέβαια, εάν θέλει κανεί να ερμηνεύσει τι συνθήκε, πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει αυτόματος σύνδεσμος μεταξύ των αποφάσεων που έχουν διατυπώσει οι πολιτικές ομάδες και της αποφάσεως που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και πιο σημαντικό ακόμη, νομίζω ότι καμία κομματική οικογένεια στις επόμενες εκλογές δεν θα μπορεί από μόνη της να συλλέξει επαρκή αριθμό εδρών ώστε να εξασφαλίσει την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα θα εξαρτηθούν όλα από τις συμμαχίες που θα αναπτυχθούν μετά τις ευρωεκλογές, ιδίως δε στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβουλεύσεως που προβλέπουν οι συνθήκες και που πιθανότατα θα γίνουν υπό τη διεύθυνση του νυν Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και που ελπίζω θα αποτελέσουν προηγούμενο και για το μέλλον. Θα είναι λοιπόν συναρπαστικές όλες αυτές οι εξελίξεις και από την άλλη μεριά πολύ ευαίσθητες. Να δούμε δηλαδή ποιο θα είναι το πολιτικό σκηνικό για τις ε, διαβουλεύσεις αυτές, καθώς επίσης ποια θα είναι η εκβασή τους. Και πρώτα-πρώτα θα υπάρξει κοινό υποψήφιο που να υποστηριχτεί από τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε αυτές να φτιάξουν ένα επαρκώς ευρύ συνασπισμό για να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες έδρες για να μπορέσει να εκλεχθεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ή για να το πω αλλιώς, οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν τον μέλλοντα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές λοιπόν θα γίνουν απόλυτα ξεχωριστά από τις παράλληλες διαπραγματεύσεις που συνήθως βέβαια διεξάγονται ταυτόχρονα για άλλα πολιτικά αξιώματα, όπως για παράδειγμα αντιπρόεδρο της Επιτροπής και είπατε εκπρόσωπο ή τον πρόεδρο του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο λίγη στα τέλη του 2014 ή για ενδεχόμενα ένα διερκή πρόεδρο του, της Ευρωομάδας, της Ευρωζώνης. Έχετε δει και εσείς πόσο δύσκολες είναι οι ισορροπίες σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η ισορροπία μεταξύ των ε, ε, φίλων, βορράς νότος, μεγάλες μικρές χώρες, ε, δύση ανατολή, διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις. Και μάλιστα, αν κοιτάξουμε και προς το παρελθόν, ενδέχεται να δούμε να υπάρξουν και πολιτικές ομάδες που να μην συμπίπτουν, για πολιτική μάλλον πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που να μην συμπίπτει με τις πολιτικές πλειοψηφίες όπως αυτές διαμορφώνονται από τις κυβερνήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βεβαίω η εκλογή του Πρόεδρου τη θα εξαρτάται από την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και αυτήν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το ειδικότερο αυτό πολιτικό περιβάλλον θα πρέπει να ανταποκρίνεται και στη διπλή φύση της Ένωσης. Ένωση πολιτών αλλά και ένωση κρατών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πιθανότατα η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βασίζεται σε κάτι σαν ένα ευρύ συνασπισμό, ένα μεγάλο συνασπισμό, που στον οποίο θα συμμετέχουν τρεις ή παραπάνω ε, κομματικές οικογένειες και εγώ προβλέπω ότι θα δούμε ε, καταστάσεις όπως αυτές που βλέπουμε και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Τέλος πάντων, για να ολοκληρώνω τώρα, πολλά θα ξεκινήσουν από τις αφετηρίες από τι οποίε θα ξεκινήσουν στις πολιτικές διαπραγματεύσεις ε, οι πολιτικές ομάδες αλλά και οι χώρες μέλη. καθώς επίσης στην ετοιμότητα των δίκαιο χαρακτήρα δηλαδή των διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν αμέσως μετά από τις ευρωεκλογέ. Και νομίζω ότι Κοινοβούλιο και Συμβούλιο είναι ίσα, εντό εισαγωγικών καταδικασμένα να καταλήξουν σε ε, συμφωνία. Δεύτερο τώρα για την πολιτική αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατά τη γνώμη μου και μιλώντας ως ιστορικός το πολιτικό έργο της Επιτροπής έγκυται πάντοτε στη συλλογικότητα και βεβαίως και το μέγεθος της Κομισιόν και στην εσωτερική της δομή. Το πολιτικό στυλ ορισμένων από τους βασικούς φορείς έχουν, έχει μειώσει την ε, εφαρμογή της αρχής της συλλογικότητας της αποφάσης της Κομισιόν. Εγώ τα έχω ξανασυζητήσει τα πράγματα αυτά και πριν από τη συνθήκη της Νίκαιας το 2000 Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ μιας ευρύτερης κομισιόν αλλά και υπέρ μιας περιορισμένης. Δεν υπάρχει βεβαίως η βέλτιστη λύση, αλλά χρειάζεται κανείς να κάνει μια πολιτική επιλογή. Η συνήθεια της Αβώνας έκανε μια πολιτική επιλογή υπέρ μιας μειωμένης αριθμητικά επιτροπής. Όμως, μετά από το Ιρλανδικό δημοψήφισμα ανατράπηκε αυτό και κατά πάσα πιθανότητα η επόμενη ε, επιτροπή θα είναι πάλι μια ευρία επιτροπή με ένα επίτροπο αναχώρα μέλος. Για να γίνει τώρα πιο συνεκτική και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να γίνει ένα είδος κορεπέρ 3, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Η πρώτη θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός συνόλου ομάδων επιτρόπων υπό την ηγεσία αντιπροέδρου εκάστοτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ενταθεί ο συλλογικό χαρακτήρα των αποφάσεων στην καθημερινή εργασία. Για παράδειγμα, ομάδα εξωτερικών υποθέσεων, ανάπτυξης, ανθρωπιστικών, αλλά και άλλες ομάδες που μπορούν να δημιουργηθούν, όπως για παράδειγμα με κύριο στόχο την ενιαία αγορά, άλλη οικονομικά και νομισματικά, τρίτη για την ε, ε, ηθαγένεια, Νομίζω η ιδέα αυτή των κλάστερ των ομάδων θα ενισχύσει τον συλλογικό χαρακτήρα της Κομισιόν. Επίσης, σε έναν αριθμό χαρτοφυλακίων, κάποιοι επίτροποι μπορούν να, λάβουν, να αναλάβουν πιο συγκεκριμένους τομείς πολιτικής που να συνδέονται άμεσα με το χαρτοφυλάκιο αντιπροέδρου ή άλλου επιτρόπου. Κλασικό παράδειγμα, ένας για τις ε, οικονομικές υπηρεσίες, που θα συνδέεται με το χαρτοφυλάκιο του ε, Επιτρόπου που έχει αναλάβει την ενιαία αγορά. Και εγώ λέω μάλιστα να είναι και αντιπρόεδρος αυτός. Οι πολιτικές αποφάσεις βέβαια όταν θα φτάσουμε στις policy guidelines αλλά και στα νομοθετικά και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες αυτές οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το σύνολο του συλλογικού οργάνου επιτροπή. Δηλαδή 28 ψήφοι και βεβαίως μία ψήφος κατά αναπρόσωπο one man, one vote ή one woman, one vote. Και ε, βεβαίως εκεί πρέπει να παίξει ρόλο και η ε, θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής για την επιλογή των διαφόρων επιτρόπων. Θα είναι δύσκολο να βρεθεί η σωστή εσωτερική ισορροπία σε ένα όργανο 28 ε, μελών, σε ένα όργανο συνολικά 28 μελών, εάν δεν έχει λέγει ο Πρόεδρος εφόσον οι χώρες μέλη προτείνουν υποψηφίους επιτρόπους για καθαρά πολιτικούς, εθνικούς στόχους και δεν λαμβάνουν υπόψη το γενικότερο ευρωπαϊκό συμφέρον, θα πρέπει οι χώρες μέλη να αναγνωρίσουν στον νέο πρόεδρο της Κομισιόν διευρυμένο περιθώριο ελιγμών και να αναγνωρίσουν ότι πολιτικά μιλώντας είναι δικαιολογημένο ο πρόεδρος της Επιτροπής να λάβει υπόψη του όχι μόνο τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα αποτελέσματα άρα, των Ευρωπαϊκών στο εθνικό επίπεδο. Θα ολοκληρώσω τώρα αναφερόμενος στην συνεργασία και στις νομοθετικές εξουσίες. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει δημιουργήσει ένα πιο ορθό, πιο ολοκληρωμένο σύστημα, νομοθετικό σύστημα δύο σωμάτων που συνεργάζονται ισότιμα. Η εμπειρία του Κοινοβουλίου από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της αγώνας αποδεικνύει ότι αυτή η προσέγγιση είναι ορθή και αποτελεσματική. Τούτου λεχθέντος οφείλει κανείς να αναγνωρίσει βέβαια ότι ότι στη διάρκεια των ετών αυτών από την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη μεταξύ ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στην άσκηση των νομοθετικών εξουσιών η Κομισιόν έχει χάσει κάποιο έδαφος. Και είναι πια ένας απλός διαμεσολαβητής. Αυτό φαίνεται και από τον αριθμό προτάσεων που αναγκάστηκε να αποσύρει η Κομισιόν, πολύ λίγο στον αριθμό. Εγώ βρίσκω ότι είναι φυσιολογική εξέλιξη αυτή. Και είναι συνέπεια της ορίμανσης του συστήματος, του νομοθετικού συστήματος των δύο σωμάτων. Παρόλα αυτά, εγώ τάσομαι απολύτως και απευθύνω έκκληση να διατηρηθεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Κομισιόν και μέσα στην εξέλιξη του συστήματος στο μέλλον. Αυτή η ισορροπία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων είναι ουσιώδη και πρέπει να διατηρηθεί ω έχει, σύμφωνα με τις συνθήκες της Αβώνα. Όπω είπε πριν ο Παύλο Ραντζέλ, θα είναι σωστό ένα τριμερές θεσμικό σύστημα να μπορεί να διευκρινίσει τα κριτήρια της νομοθεσίας των κατεξουσιοδότης πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Διάκριση που είναι πρόσφατη γιατί την έφερε σε φως η συνθήκη της Λεσαβόνας και είναι θεμελιώδες να συμφωνήσουν τα τρία θεσμικά όργανα για τα κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμόζονται, να χρησιμοποιούνται και να εφαρμόζονται όταν συντάσσεται η νομοθεσία, όταν ασκούνται οι νομοθετικές ουσίες και βεβαίως ποιος, ποιο είναι πραγματικά το πεδίο εφαρμογής των πράξεων αυτών, των κατά εξουσιοδότηση πράξεων. Γνωρίζω ότι είναι απαραίτητο να συνδυαστεί συνεργασία μεταξύ των, των, θεσμών και βεβαίως και τα ετήσια και πολιετή προγράμματα εργασιών, αλλά και οι διαθεσμικές συμφωνίες, οι οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνουν δεχτές από τα τρία θεσμικά όργανα ως τέτοια αποφεύγοντας έτσι άλλες επιμέρους διαθεσμικές ε, συνεργασίες που μπορούν να αποδειχτούν αντιφατικές και πάντως δεν θα συμβάλλουν στο ξεκαθάρισμα των πολιτικών στόχων του συνόλου της Ένωσης. Ενώ πιστεύω ότι η σαφήνεια στόχων ακριβώς είναι κάτι που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα, κυρίε και κύριοι, έτσι ώστε το 2014 να αποτελέσει το εφαλτήριο για την συμφιλίωση των πολιτών μας, της πλειοψηφίας των πολιτών μας με το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Ευχαριστώ τον καθηγητή Βιτορίνο. Επανέρχομαι στο θέμα της έκθεσης και στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και μετά θα μιλήσουν οι υπόλοιποι βουλευτές μέχρι τις 4.30. Σεπλίν. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, μια στιγμή προσεξίας. Δεν άκουσα. Συγγνώμη, θα αρχίσω τώρα. Ε, το θέμα που συζητούμε νομίζω είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Έχει κεντρική σημασία για τη μελλοντική πορεία της Ένωσης και ο Πάλο Ράντζελ ε, έκανε πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις ε, από αυτού. Εγώ θεωρώ ότι και θα καταλάβετε σε λίγο για ποιο πράγμα μιλώ. Το πρόβλημα είναι το 2005 και τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και την Ολλανδία. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα. Η φθήνουσα υποστήριξη από πλευράς του λαού για το ευρωπαϊκό εγχείρημα που ε, συνοδεύει την ευθύνουσα νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, αλλά πάντως νομίζω ότι ε, αυτή είναι η πηγή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Όλοι είμαστε προσιλωμένοι στην δημοκρατία, στο δημοκρατικό σύστημα, αλλά υπάρχει το εξής παράδοξο, δεν υπάρχει ταύτιση ε, με το ευρωπαϊκό δημοκρατικό οικοδόμημα και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις χώρες που γνωρίζω πολύ καλά αυτό διαπιστώνω. υπάρχουν διάφορες προτάσεις από πλευράς ε, του κυρίου Ραγκέλ για να υπερπηδήσουμε αυτές τις δυσκολίες. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Ε, μίλησε για το διαχωρισμό των εξουσιών. Δίκιο έχει. Όταν ε, μιλάμε για δημοκρατία είναι κεντρική σημασία ο διαχωρισμός των εξουσιών. Αυτή τη στιγμή σε επιτευχθεί ο διαχωρισμός θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι διαδικασίες σε σχέση ε, με το πώς θα διασυνδέω τα διάφορα τεμήματα της ε, κυβέρνησης ή διακυβέρνησης, να το πω καλύτερα. Νομίζω ότι ε, παρότι έχει ε, σημειωθεί πρόοδος, ε, δεν έχουμε επιτύχει το στόχο μας σε σχέση με την μη άμεση εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά πάντως αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος μας ο τελικός στόχος μας. Στη συνέχεια, οι υποψήφοι επίτροποι, πιστεύουμε, ε, βάσει της πρότασης μάλλον του κυρίου Ραγκέλ, θα πρέπει να ε, προέρχονται από ε, τους ευρωβουλευτές. Νομίζω ότι έτσι θα δημιουργηθεί ένα υβριδικό σύστημα που δεν με βρίσκει σύμφωνο, διότι θα ψηφίζουν για τους εαυτούς τους και στη συνέχεια θα ψηφίζουν για να βγει ο πρόεδρος, για να καταλάβουν τη θέση του επιτρόπου. Νομίζω ότι θα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα νομιμοποίησης ε, στη συνέχεια και κυρίως σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Ως προς το ρόλο των εθνικών ε, κοινοβουλίων, είτε μας αρέσει είτε όχι, απολάβουν μεγαλύτερες νομιμοποίηση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω το ρόλο τους και τις μελλοντικές τους αρμοδιότητες ε, στα πλαίσια της ε, νέας θεσμικής αρχιτεκτονικής. Πιστεύω σε κάθε περίπτωση ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενισχυθεί. Εγώ παρατηρώ ότι στις ε, Βρυξέλλες έχει συγκεντρωθεί ε, υπερβολικά μεγάλη εξουσία και υπερβολικά πολλές αρμοδιότητες στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μεγάλη απόσταση από τους ε, πολίτες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε πραγματικό δήμο πλέον και άρα δεν μπορούμε να έχουμε ουσιαστική δημοκρατία με την οποία θα ταυτιστεί ο λαός. Ίσως θα έπρεπε να εμφανίζεται και να λογοδοτεί και στα Εθνικά Κοινοβούλια ο Πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, η πρόταση για τους Επιτρόπους άνευ χαρτοφυλακίου ίσως είναι μία οδός, αλλά δεν καταλαβαίνω. Οι άνευ χαρτοφυλακίου Επίτροποι τι ακριβώς θα κάνουν. Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων είναι υποσυζήτηση το ζήτημα. Αναρωτιέμαι αν ε, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, για το νομοθετικό έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα Εθνικά Κοινοβούλια. Νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε σοβαρές συγκρούσεις συμφερόντων. Πιστεύω ε, πως χρειαζόμαστε επίσης μια πολύ πιο αποτελεσματική επικοινωνιακή πολιτική. Η πολιτική μας μέχρι τούδε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, η αποτελεσματικότητά της ε, βλέπουμε ε, ότι έχει πάρα πολύ συχνά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Εάν πάτε στην ε, Ουγγαρία και ρωτήσετε ε, τους περαστικούς ποιος είναι ο επίτροπός σας, ε, η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα έχει ιδέα. Δεν είναι καλό αυτό. πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα σε αυτό ακριβώς το τομέα το 2004 δρομολόγησε μια νέα επικοινωνιακή πολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την προηγούμενη θητή, αλλά τελικά εξέλιψε, εξαφανίστηκε, εξανεμίστηκε. Δεν ξέρω τι έγινε. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα. Δεν είναι εύκολο. Ε, υπάρχει συγκεντρωμένη εξουσία στις ε, πολιτικού χαρακτήρα, μεταμφιεσμένη ως τεχνοκρατική ενίοτε, αλλά σε κάθε περίπτωση τα ΜΜΕ θα πρέπει να αναμεταδίδουν τι πληροφορίε. Ξέρουμε ότι δεν είναι και τέλεια. Σε κάθε περίπτωση κάτι μπορούμε να κάνουμε ε, με τρόπο ώστε να καλύψουμε τουλάχιστον ένα μέρος ε, του χάσματος ε, που υπάρχει ανάμεσα στην Ένωση και του πολίτε τη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω υπόλοιπα μέλη τη Επιτροπής και του συντονιστέ να ολοκληρώσουν παρακαλώ και μετά θα επιστρέψουμε στους κύριους ομιλητές. Ο κύριος Λάινεν έχει ζητήσει το λόγο για τη σοσιαλιστική ομάδα αντικαθιστά τον υπεύθυνο της αντιπροσωπείας τον κύριο Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Πάουλο Ραουζέλ για την σημαντική έκθεση που θα κληθούμε να ψηφίσουμε άλλωστε σύντομα καθώς και τον Αντώνιο Βιτορίνο προς τον οποίο απευθύνω χαιρετισμό και ο οποίος ανέπτυξε ορισμένες χρήσιμες ιδέες για την ε, για το εναρκτήριο λάκτισμα. Όμως η συνθήκη της Λισαβόνας που είχε αποτελέσει ε, αντικείμενο μακρότατων διαπραγματεύσεων στη συνθήκη, στην συνέλευση τότε, είχε πει ότι η συνθήκη λέει ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι προεδρική. Η προεδρευόμενη. Επομένως, ο πρόεδρος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκλέγεται όχι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πλέον όπω το παρελθόν, αλλά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα σημαντικό βήμα προ τον εκδημοκρατισμό τη Ευρώπη, δυνάμει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και επειδή τώρα προτίθεται, προτίθεμεθα μάλλον να κάνουμε, να δούμε πώ θα λειτουργήσει, γι' αυτό εγώ προειδοποιώ προσοχή, να μην αρχίσουμε να σκεφτόμαστε άλλες εναλλακτικέ μεθόδους, ίσως και την απευθείας εκλογή του Προέδρου της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι που είχε και λίγο λαϊκιστικά. Είχε συζητηθεί τότε πολύ. Απερίφθη εν τέλει από τις 28 αυτές χώρες με τα πολύ διαφορετικά συμφέροντα η κοινοβουλευτική διαδικασία που είναι σημαντικότερη για να δεσμεύονται και τα κόμματα και για να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση και με τις τοπικές κοινωνίες, κοινότητες, περιφέρειες κτλ. Ενώ οι ευρωεκλογέ θα είναι η αρχή της θεσμοποίησης. Δεν μπαίνει στο σύστημα. Και Παύλο, ελπίζω στην έκθεσή μας να το αφαιρέσουμε αυτό, διότι είναι απολύτως εκτός τόπου και χρόνου να αρχίσουμε να οικοτολογούμε, όπως κάνουν ορισμένοι που δεν τους έρχεται καμιά καλύτερη ιδέα και στην χώρα μου, την Γερμανία, καμιά φορά πέφτει αυτό σαν αλεξιπτότης ως ιδέα δηλαδή. Η ιδέα της εκλογής του, του... Της εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τόσο ισχυρή που δεν πρέπει να την αμφισβητούμε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έτσι θα γίνει κιόλα τον Ιούνιο. Και η καγκελάριος μου είπε ότι δεν είναι αυτόματος ο σύνδεσμος. Όχι, έτσι είπε. Είναι όμως αυτόματος ο σύνδεσμος. Εφόσον θα έχουμε εμείς εκλέξει, θα γίνουν διαβουλεύσεις, θα γίνουν διαπραγματεύσεις, θα διαμορφωθούν πλειοψηφίες στο Κοινοβούλιο και σύμφωνα με αυτές τις διαμορφούμενες πολιτικές πλειοψηφίες θα κληθεί να κάνει πρόταση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ τίνω, όπως και πολλοί από τους φίλους μου, να μην ψηφίσω κανένα από τους προταθισόμενους, εφόσον αυτό το πρόσωπο δεν υπήρξε ε, υποψήφιος σε ευρωεκλογέ. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας αυτόματος χαρακτήρας εδώ στην διασύνδεση αυτή. Είπε ο Βιτορίνο ότι θα φτιαχτούν πακέτα, θα φτιαχτεί ένα πακέτο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί με τα άλλα υψηλά αξιώματα όπω ε, την είπα τη εκπρόσωπο για τι εξωτερικέ σχέσει, τον ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. όμω εδώ κάνουμε σύγκριση ανώμιων πραγμάτων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό. Άλλο η πρόταση για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να προκύψει μέσα από τις ευρωεκλογέ. Εγώ νομίζω ότι το Κοινοβούλιο κατέκτησε την ε, συναπόφαση μέσω της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας και πράγματι λόγω της κρίσεως υπήρξε και κάποια μετακίνηση από την κοινοτική μέθοδο στην διακυβερνητική. Κάτι το οποίο πρέπει να επαναφέρουμε στο σωστό δρόμο. Στην άλλη έκθεση Είπαμε τι θέλουμε. Θέλουμε να εξαντλήσουμε την συνθήκη. Η Επιτροπή έχει πολύ μεγαλύτερες εξουσίες από αυτές που χρησιμοποίησε ως Επιτροπή Μπαρόσο 2. Υπάρχουν ακόμα εξουσίες που δεν τις έχει εξαντλήσει, δεν τις έχει χρησιμοποιήσει και εκεί στα κενά που άφησε η αδράνεια της αυτή έτρεξαν και μπήκαν οι χώρες μέλη. δεν έχουν χώρο εδώ εξωκοινωτικέ διαδικασίες. Εμείς έχουμε ορισμένες επιθυμίες για τον εκδημοκρατισμό και το δικαίωμα πρωτοβουλία είναι δικαίωμα υπαρξιακό κάθε βουλής. Έχουμε καλύψει ένα μέρος του δρόμου, να αντιδρά δηλαδή η Κομισιόν σε εκτιθέμενες ε, επιθυμίες του Κοινοβουλίου, αλλά ακόμα δεν έχει κατακτηθεί όλο το όλον εφόσον έχει εκφραστεί το Κοινοβούλιο με σαφέ αποτέλεσμα σε πλειοψηφία στην ολομέλειά του, τότε πρέπει να αντιδράσει η Κομισιόν με κατάθεση νομοθετικής προτάσεως ώστε έχουμε σχεδόν δίκαιο πρωτοβουλία. Όχι μεν τυπικό, αλλά ουσιώδε, εφόσον αντιδρά σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέλευση, αγαπητέ Βιτορίνο, είχαμε συζητήσει διαμακρών το ενδεχόμενο η Κομισιόν να είναι μικρότερη διότι αν κάποια στιγμή μπουν όλες οι συνιστώσεις της πρώην Ιουκοσλαβίας θα έχουμε 35 επιτρόπους. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει καλά το σύστημα αυτό. Ίσως λοιπόν όχι τώρα, αλλά την επόμενη φορά κάτι πρέπει να γίνει. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι στην νυν έκθεσή μας δεν θα πρέπει να θέσουμε θέμα αριθμού επιτρόπων. Θα πρέπει να εγγύψουμε περισσότερο στην εσωτερική δομή της Επιτροπής αυτή η δημιουργία των ομάδων υπό την κατεύθυνση ενός ε, αντιπροέδρου είναι μια καλή ιδέα και πιστεύω και ελπίζω ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής να δράξει την ευκαιρία και να τα εφαρμόσει τα πράγματα αυτά. Πρόεδρος της Επιτροπής που θα έχει εκλεγεί από το Κοινοβούλιο θα είναι μια προσωπική, προσωπικότητα, πολιτική προσωπικότητα μεγάλης βαρύτητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να επιβάλλει όρους ώστε να μπορεί να απορρίψει προτάσεις των εθνικών κυβερνήσεων. Έχει συμβεί αυτό, θα μπορέσει να συμβεί ακόμη περισσότερο. Τις υποψηφιότητες δηλαδή. Όταν δηλαδή απλά κάποια κυβέρνηση επιθυμεί να ξεφορτωθεί κάποιον στέλνοντάς τον στις Βρυξέλλες, να μπορεί να το απορρίψει. Ο Παύλ Ραντζέλ είπε ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον τρεις προτάσεις υποψηφιότητων. Αυτό είναι κάπως τυπολατρικό. Εγώ προτιμώ να βασιστώ την ε, ισχύ, την βαρύτητα της θέσης του νέου Προέδρου της Επιτροπής που θα μπορεί να πει όχι σε κάποιες υποψηφιότητες. Ελπίζω πολύ, Επίτροποι, να προέλθουν και από ε, εθνικές βουλές. Πολλοί θα κατέβουν υποψήφοι, κάποιοι που υπήρξαν ήδη επίτροποι θα ζητήσουν να ξαναείνε υποψήφοι, γιατί όχι, εάν ταιριάζει από άποψη σχετισμού πολιτικών δυνάμεων. Λόγω τη ε, σχετική πιέση χρόνου θα αρκεστώ σε αυτά. Ένα δικαίωμα ωστόσο που θεωρώ ότι έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη συνθήκη και που νομίζω δεν το έχει ασκήσει, είναι το δικαίωμα πρωτοβουλία για την αναθεώρηση των συνθήκων. Έχουμε πλήρωνε προτάσει όπου έχουμε διατυπώσει τις απόψεις μας σχετικά με το τι δεν πάει καλά. Ελπίζω, αν όχι τούτο το κοινοβούλιο τότε το επόμενο, να χρησιμοποιήσει το διενές προνόμιό του για να συγκαλέσει νέα συνέλευση και να δώσει νέα όθηση, νέα κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόσμος σιγά σιγά μπαίνει στα στασιμότητα, η Ευρώπη μπαίνει στα στασιμότητα, χρειαζόμαστε κάποια νέα όθηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Λάινεν. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Νταφ, να χαιρετήσω τον κύριο Ρος, ο οποίος θα πάρει για πρώτη φορά το λόγο σε λίγο αντικοθιστώντας τον συνάδελφο Τραϊκόσκι. Είναι πρώτη φορά που είναι εδώ και τον συγχαίρω. Δίνω το λόγο στον κύριο Νταφ. Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίζω και εγώ τον Αντώνιο Βιτορίνο. Είναι καλό να βλέπει κανείς τους παλαιούς της ε, Σύμβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την συνέλευση μάλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν πράγματι έχει υπάρξει πρόοδος και θα πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ήταν ένα θετικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκάλεσε σημαντικά βήματα προόδου για την δημοκρατία και εκεί που δεν προχώρησαν τα πράγματα είναι στο ότι δεν δημιουργήθηκε μια σωστά προσιλωμένη θα έλεγα και ισχυρή εκτελεστική εξουσία. Εγώ νομίζω ότι δεν λείπει το Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κυβέρνηση. Δεν μπορεί κανένας να θέλει ισχυρότερο Κοινοβούλιο αν δεν έχει ισχυρότερη κυβέρνηση η οποία θα αντιδρά και θα αλληλοεπιδρά. Τα επόμενα πέντε χρόνια θα πρέπει να ληφθεί μια κρίσιμη, μια ιστορική απόφαση για όλους. Θα δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την αρμοδιότητα να είναι ο πυρήνας της εκτελεστικής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας τις εξωτερικές υπηρεσίες για να θέσει σε εφαρμογή τις δράσεις και να χρησιμοποιεί την, γραμματεία σαν, την Επιτροπή συγγνώμη, σαν ένα είδος γραμματείας. Αυτή η επιλογή φαίνεται ότι προωθείται και από την Καγκελάριο η οποία θέλει να ξεπεράσει το πλαίσιο το κοινοτικό. Όπως μας είχε πει στην ομιλία της στην Μπρίζ, να προχωρήσει στην εφαρμογή της λεγόμενης κοινοτικής μεθόδου ή εννοσία μεθόδου. Μια δεύτερη επιλογή, η οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι και πιο πιθανή να συγκεντρώσει τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών και των κοινοβουλίων των κρατών μελών Η εναλλακτική λύση βέβαια είναι το αντίθετο, είναι η ομοσπονδιακή λύση. Να προσπαθήσουμε να κρατηθούμε στο εσωτερικό της συνθήκης να προσφύγουμε στην μεγαλύτερη δυνατή χρήση της μεθόδου Μονέ, όπου αυτό είναι εφικτό, και να μετασχηματίσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι είναι σήμερα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά να την μετατρέψουμε από αυτό που είναι σε, σε μια πραγματική ουσιαστική ε, κοινοβουλευτικού τύπου κυβέρνηση. Τώρα οι διαδικασίες αυτές όλες με τους σκιώδεις υποψηφίους και τα λοιπά μέχρι τώρα δεν έχουν αποδώσει. Και θα επηρεάσουν άλλωστε κατά πολύ την έκβαση ε, της προσπάθειας την οποία αναλαμβάνουμε και της επιλογής την οποία θα πρέπει να κάνουμε. Η εμπειρία αυτή είναι ένα πείραμα. Ε, μπορεί και να αποτύχει αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και γι' αυτό υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Στοιχεία τα οποία στην παρούσα στιγμή δεν φαίνεται να εκτίθενται στον τύπο και να φαίνονται ότι είναι παρόντα στην κοινοβουλευτική συζήτηση. Ο προτινόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνει γνωστός τον μήνα Ιούλιο από ό,τι φαίνεται, ίσως και τον Αύγουστο. Αυτή η επιπλέον νομιμοποίηση από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο θα οδηγήσει το πρόσωπο αυτό στο να αφήσει σφαγίδα, τη σφαγίδα του ε, στο νέο σύνολο των επιτρόπων. Θα έχει δηλαδή το ειδικό βάρος, την εμβέλεια, τις πολιτικές απόψεις Ο κύριος Βιτορίνου αναφέρθηκε σε τέτοιες υποθέσεις. Αλλά δεν θα γνωρίζουμε αν το πείραμα αυτό θα πετύχει πριν δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα και ποιος είναι ο νέος προτινόμενος πρόεδρος ο οποίος θα πρέπει να αρνηθεί να είναι σε θέση να αρνηθεί και τον προτινόμενο ορισμό ενός επιτρόπου αν δεν του κάνει. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το πώς θα επηρεάσουν οι αλλαγές αυτές την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στάθηκε ικανό να αποκτήσει θα έλεγα αρκετές αρμοδιότητες τις οποίες η συνθήκη δεν καθορίζει και δεν προβλέπει με αυστηρό τρόπο. Καλείται το Συμβούλιο όμως να αναλάβει και μια υψηλή σημασία συνταγματική αποστολή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή but not before the Καταρχάς θα προτείνει το σχηματισμό της Επιτροπής ε, στις αρχές Ιουλίου και όχι νωρίτερα θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το νέο κοινοβούλιο να, διαβολη, να διαβουλευτεί με αυτό και να ζητήσει τον σχηματισμό της ε, νέας επιτροπής. για αυτούς οι οποίοι πιθανώς αμφισβητούν το θεσμικό, το κρατικό, αν θέλετε, την κρατική υπόσταση της κοινοτικής πολιτικής, προσέξτε, γιατί μπορεί να δημιουργήσετε ε, μια θέση η οποία να έχει τόσες πολλές αρμοδιότητες που θα μειώσει ε, την κοινοβουλευτική αντιστάθμιση που είναι απαραίτητη στη δημοκρατία. Τίθεται και αυτό σαν ερώτημα. Τρίτον, τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τα οποία υποτίθεται θα ορίσουν και στη συνέχεια θα στηρίξουν μέσω μιας ιδιαίτερως πολλωμένης πολιτικής αντιπαράθεσης, προεκλογικής αντιπαράθεσης τους υποψηφίους τους. Είναι σαφές ότι για αρισμένα από τα πολιτικά κόμματα κάτι τέτοιο ήδη στην παρούσα φάση δοκιμάζει την ενότητά τους και την οργανωτική τους ακαιρεότητα και κατεύθυνση. Η φιλελεύθερη ομάδα, της οποίας είμαι ευτυχές μέλος, αντιμετωπίζει σημαντικότατες ανταγωνιστικές θα έλεγα καταστάσεις ανάμεσα σε δύο ισχυρά φιλελεύθερα στελέχη που εκπροσωπούν τις δύο πλευρές αν θέλετε της ε, κρίσιμης επιλογής την οποία κατέθεσα στην αρχή της παρουσίασής μου η φεντεραλιστική άποψη η οποία εκπροσωπείται από τον Φερχόφστατ. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα βγει από την αντιπαράθεση αυτή η φιλελεύθερη ομάδα. Αλλά πάντως θα έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για μας νομίζω αλλά και για τον μελλοντικό προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φερχόστατ από τη μία, η επιλογή των Γερμανών και της Μέρκελ από την άλλη. Λόγω ακριβώς της σημαντικής θέσης που έχει η ομάδα των φιλελευθέρων στο σώμα αυτό και ο ρόλος μοχλού που μπορούν να παίξουν. Ε, οι σοσιαλιστές θα επιλέξουν έναν υποψήφιο από έναν υποψήφιο, κάτι το οποίο τους αρκεί. Οι πράσινοι ε, θα περάσουν από εσωκομματικές εκλογές, καλή διασκέδαση και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει πολλούς πρωθυπουργούς, τέος πρωθυπουργούς, υποτιθέμενους πρωθυπουργούς, πιθανούς πρωθυπουργούς που όλοι αυτοί θα ήθελαν τη θέση. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί με αυτούς τον Μάρτιο. Δεν ξέρω α, πώς θα λειτουργήσουν τα πολιτικά κόμματα, αν θα επιβιώσουν από αυτή τη διαδικασία ή αν θα διασπαστούν. Πάντως για το Κοινοβούλιο ο μαγικός αριθμός είναι 376, 376 ψήφοι. Ο αριθμός των μελών δηλαδή που θα πρέπει να στηρίξουν ένα ή οδήποτε εκπρόσωπο ο οποίος θέλει να έχει πιθανότητες επιτυχίας και να προεδρεύσει σε κάποια φάση της Επιτροπής. Κοιτάξτε, μακρηγόρησα και θα σταματήσω εδώ. Θα είχα πολλά να πω επίσης και για το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είμαι βέβαιος όπως ο κύριος Βιτορίνο ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση καλύτερη βέλτιστη λύση. Αλλά εγώ έχω κάποιες προτάσεις τις οποίες θα χαρακτήριζα μάλλον και δραστικές. Ευχαριστώ κύριε Νταφ. Ο συνήθως η παρουσίασή σας είναι πλήρης νοημάτων και δίνω αμέσως το λόγο στον συνάδελφο Φόξ. Ευχαριστώ. Πολύ χαίρομαι που μιλώ μετά τον Άντριο Ντάφ ε, από τον ίδιο συνασπισμό. Ε, κάποιοι ξέρουν ε, ότι έχουμε υιοθετήσει μάλλον διαφορετικές απόψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Βιτορίνο και τον κύριο Ράγκελ για τις παρουσιάσεις τους. Μιλήσαμε πολύ για έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε για την έλλειψη της νομιμοποίησης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι Επιτροπή ε, εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι όπως άρχισε έτσι και εξακολουθεί να είναι μια ένωση εθνικών κρατών που βασίζονται σε διεθνικές ε, συνθήκες. Ε, τα τελευταία χρόνια έγινε μια απόπειρα τροποποίηση των συνθήκων και είχαν το θάρρος κάποιοι λαοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το αρνηθούν. Αν, ήμασταν, αν ήταν δημοκρατικό το σύστημα θα το είχαμε δεχθεί. Όμως τι γίνεται, επανέρχονται οι ίδιες συνθήκες υπό διαφορετική μορφή. Αν είστε από την Ιρλανδία και την Δανία, μικρή δηλαδή σας λένε ξαναψηφίστε ε, και ε, ότι περίεργο είναι καταφατική απάντηση στη συνέχεια και αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα αλλάξει ο τίτλος της συνθήκης ε, και ε, θα, αντί να μιλάμε για σύνταγμα θα το ονομάζουμε συνθήκη της Λισαβόνας αλλά το 85% του DNA είναι το ίδιο ακριβώς. Θλίβομαι που επικυρώθηκε από την Βρετανία το, η συνθήκη της Λισαβόνας προτού καν μας δοθεί η, η ευκαιρία να αποφανθούμε κι εμείς σε ένα δημοψήφισμα, διότι ε, ένα πολύ μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων εκχωρούνται από το Westminster ε, στις Βρυξέλλες ε, χωρίς τη συγκατάθεση του λαού. So I don't regard the EU as terribly democratic at... Ε, πάντως ε, δεν είναι καθόλου δημοκρατικό αυτό το σύστημα, ούτε και το ίδιο το κοινοβούλιο δεν είναι δημοκρατικό. Στι εκλογές που διεξάγονται πολύ λίγοι μετέχουν ε, και όταν συμμετέχουν ουσιαστικά είναι μία για κατά των εθνικών κυβερνήσεων. Εμείς οι πολιτικοί ξέρουμε ότι αυτό ισχύει. Είπε ο κύριος Φλίνγκ ότι αν ζητούσε από τους ψηφοφόρου του να κατονομάσουν τον Ευρωπαίο Επίτροπο, πολύ λίγοι θα ε, ήξερα να το κάνουν το 2%. 2%. Πολύ ενδιαφέρον ποσοστό γιατί το ίδιο ισχύει και για τους Βρετανούς ψηφοφόρους ε, όταν τους ρωτάμε ποιοι είναι οι ευρωβουλευτές σας. Ε, τα εθνικά κοινοβούλια αντίθετα έχουν ένα 50% και βλέπουμε ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη νομιμοποίηση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα ε, θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία τη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με υπουργού ε, που ε, μπορούν να αποπευθούν από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό θα ήταν η λύση. Και αν θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερο έλεγχο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ενισχύσουμε τη διαδικασία τη κίτρινη κάρτα που εισήχθη στην συνθήκη τη Λισαβόνα. δυσχρησιμοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε και προ το παρόν έχει απλώ αγνοηθεί για την διαδικασία της κίτρινης ε, κάρτας ε, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να τροποποιηθεί θα πρέπει να απαιτούμε μόνο τρία και όχι εννέα εθνικά κοινοβούλια για τη σύμφωνη γνώμη τους για να εκκινήσει αυτή ε, η διαδικασία της ε, ε, γίτρινη κάρτα και να ξανασκεφτεί κάποιο ζήτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συντακτική συνέλευση θέλησαν να δημιουργήσουν την ψευδέστηση της συγκρότηση ενός νέου μηχανισμού καθιστώντα όμως αδύνατη την ε, ε, λειτουργία αυτού του μηχανισμού. Ο κύριος Λάινεν ε, μας είπε ότι λυπάται πως το Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 48 δεν έχει εισηγηθεί οποιασδήποτε ε, τροποποιήσεις στη, για τη συνθήκη. Δεν προσπαθήσαμε, το δική σας ομάδα παρεμπόδισε το, τη δική μας προσπάθεια, τη δική μου πιο συγκεκριμένα, να έχουμε μία έδρα για να εκπροσωπείται και το Κοινοβούλιο. μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία, το 75 ε, των βουλευτών θέλει να έχει μία έδρα μόνο το Κοινοβούλιο ε, και εσείς ε, και η ηγεσία του Κοινοβουλίου και κλεισμένο των θυρών παρεμπόδισαν αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα θα επανέλθει αυτό στην επόμενη θητεία. Ξέρετε όμως ότι... Δεν δικαιούστε να δηλώνετε ότι ε, θλίβεστε για την ε, έλλειψη τροποποιήσεων. Γιατί δεν μιλάτε με τον κύριο Σβόμποντα ή με τον κύριο Γουαλτιέρη ε, και να, τους, να μας εξηγήσουν γιατί δεν επιτρέπουν τροποποίηση της συνθήκης βάσει του άρθρου 48. Τι πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε την νομιμοποίηση. Ας κάνουν ό,τι κάνανε πάντοτε τα εθνικά κοινοβούλια, δηλαδή να ζητήσουν να λογοδοτήσει το εκτελεστικό όργανο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει λογοδοσία για τις δαπάνες κανονικά. Τι βλέπουμε όμως να συμβαίνει το ελεγκτικό συνέδριο κάθε χρόνο αρνείται να ε, υπογράψει τους λογαριασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι είναι μεγάλο το ποσοστό λάθους και τι κάνουν οι βουλευτές, ε, υποψηφίζουν τους προϋπολογισμούς ούτως ή άλλως. Αυτό δεν είναι λογοδοσία και έλεγχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμμετέχουμε απλώς σε ένα φεντερελιστικό εγχείρημα. Μπορεί να συμφωνείτε όμως, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι δεν χρησιμεύει αυτό το φεντερελιστικό οικοδόμημα όταν κανείς δεν λογοδοτεί για την ε, κατασπατάληση των ε, πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να ε, λογοδοτούν οι επίτροποι, να αποπέμπονται οι επίτροποι. Το ίδιο συμβαίνει και στις επιχειρήσεις. Οι μέτοχοι διαλύουν το Διοικητικό Συμβούλιο όταν δεν μπορούν να λογοδοτήσουν για τις δαπάνες. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς με τα μέλη της Επιτροπής. Θα έπρεπε επίσης να νομοθετήσουμε Ευχαριστούμε λιγότερο, διότι όσο περισσότερο είναι ο νόμοι, τόσο δυσκολεύει το έργο των επιχειρήσεων, χάνονται και άλλε θέσει εργασία και ανταυτού θα έπρεπε να ελέγξουμε με ποιο τρόπο εφαρμόζονται τα εφιστάμενα νομοθετήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή να πω καλύτερα πω δεν εφαρμόζονται σε κάποιο μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, διότι ε, στην ε, δική μου εκλογική περιφέρεια διωγγώνεται η δυσαρέσκεια, διότι θεωρούν όλοι ότι στην Βρετανία μέχρι τελευταία τελευταίας κεραίας εφαρμόζουμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαστολή με άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματος χάρη, ε, με τα, η κλοβή, τα χειροστάσια, με το μέγεθος των κλοβών, τέτοιου είδους νομοθεσίες ε, ε, δεν εφαρμόστηκαν ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μήνες μετά την έγκρισή τους, ενώ είχαν εφαρμοστεί στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και δημιουργείται, καταλαβαίνετε, δυσαρέσκεια και θορυβείται ο λαός, διότι βλέπω δεν υπάρχει ομοιόμορφη ε, εφαρμογή. Θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ίδια. Ε, προετοιμαζόμαστε αυτή τη στιγμή για την ή ε, μία μεσή εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ ε, προσωπικά πιστεύω ότι είναι ψευδεπίγραφη και δεν νομιμοποιείται αυτή η εκλογή. Θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα. Δεν αναφέρεται πουθενά συγκεκριμένα ότι πρέπει να ορίζουν υποψηφίου στα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες και τουλάχιστον στη δική μου εκλογική περιφέρεια όταν ψηφίζουν οι ψηφοφοροί, τουλάχιστον ξέρω ότι δεν θα έχουν την παραμικρή ιδέα ποιοι θα είναι οι υποψήφοι των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων. Και πιστεύω ότι αυτό ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό είναι δικαίωμα του Συμβουλίου και δεν θέλω να ε, αλλάξουν τα πράγματα. Η δική μου πολιτική ομάδα δεν έχει ορίσει υποψήφιο ε, και νομίζω ότι με σιγουριά μπορώ να προβλέψω ότι δεν θα το κάνουμε, δεν θέλουμε να ε, συμμετάσχουμε σε αυτήν την εκλογή είναι γελίο που ε, οι σοσιαλιστές όρισαν υποψήφια από έναν τελικό κατάλογο όπου υπήρχε μόνο ένα όνομα. Ε, κύριε Ράντζελ, στην δική σας έκθεση λέτε ότι οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει εγκαίρως να ορίζουν τον υποψήφιό τους εγκαίρως πριν από τις εκλογές ε, και το ΕΛΚ δεν θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα μέχρι το Μάρτιο, δηλαδή δύο μήνες πριν τις εκλογές. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα ξέρετε ποιος είναι υποψήφιος για την Προεδρία ή ο υποψήφιο ε, για την κυβέρνηση μήνε, χρόνια νωρίτερα θα το γνωρίζατε, οπότε δεν είναι φυσιολογικό. Θεωρώ, λοιπόν, ξαναλέω, ότι είναι ε, επίπλαστη ε, αυτή η διαδικασία ψηφοφορία και θέλω να καταλάβω τι θα συμβεί αν οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε πάρουν περισσότερε έδρε από το ΕΛΚΑ και διεκδικήσουν την νίκη στι εκλογέ, αλλά παρόλα αυτά στο Συμβούλιο έχετε κεντροδεξιά πλειοψηφία υποψηφία στο Συμβούλιο, διότι μπορώ να καταλάβω πώς θα ε, ε, ε, βάλουν τον κύριο Σούλτσε με αυτή την πλειοψηφία, αλλά τέλος πάντων τα πάντα μπορεί να περιμένει κανείς τη σημερινή ημέρα. Τέλος, συμφωνώ κύριε Βιτορίνο με αυτά που μας είπατε για τα κλάστερ στις ομάδες των επιτρόπων. Θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουμε από πολιτική σκοπιά να μειώσουμε τον αριθμό των επιτρόπων, οπότε η ιδέα από τους 28, οπότε το να έχουμε αντιπροέδρους, δηλαδή ουσιαστικά υφυπουργού 6-7 το αριθμό θα ήταν μια καλή ιδέα. Δεν ξέρω η Επίτροπη ή οι υπόλοιποι Επίτροποι τι κάνουν όλη την ημέρα. Ε, τα, τελευταία 4,5 χρόνια τι κάνει ο επίτροπο ε, για τη διεύρυνση. Λίγα φαντάζομαι τις ε, για το επόμενο πρόγραμμα εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα ήθελε οι Επίτροπη να έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Παραδείγματο χάρη, θα μπορούσαμε να έχουμε για την ε, συμφωνία, την Διατλαντική Συμφωνία για τι Επενδύσει, έναν Επίτροπο που θα ασχολείται με αυτό. Ή επίση ένα άλλο να ασχολείται με τι εμπορικέ συναλλαγέ με την Κίνα. Ποια είναι, ποια η βασική μα αποστολή, να προωθήσουμε το ελεύθερο εμπόριο και να αναβαθμίσουμε την εσωτερική αγορά αγορά. Τέλος, Πρόεδρε, θα έπρεπε να ασχοληθούμε και να προσιλωθούμε στους αρχικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να αυξηθεί η ευημερία των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να δημιουργήσουμε μια πολιτική ένωση που όλοι απέφχονται, διότι κάθε φορά που τους δίνεται η ευκαιρία να το ψηφίσουν, καταψηφίζουν αυτή την πρόταση των Βρυξελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε αρχικές αποστολές, ελεύθερο εμπόριο, ενιαία αγορά, έτσι θα ενισχύσει πάρα πολύ τη φήμη της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Άγνιου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα μιλήσω για 9 λεπτά. Θα πάμε λίγο πιο γρήγορα με μένα. Ο κύριος Σόφλινγκ μίλησε για το 98% των Ούγγρων που δεν γνωρίζουν τον επίτροπό τους. Γελώ, όχι γιατί θέλω να εξυβρίσω τους Ούγκρους, αλλά να ρωτήσω και στη δική μου μικρή πόλη, μια εμπορική πόλη, ε, ποιος είναι, κανένας δεν ξέρει, άντε να θυμηθούν τον Μάντελσον ή κάποιον άλλο. Ο Φόξ μας είπε «Ε, το τι δεν πήγε καλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι εξουσίες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μα τους τη δώσανε την εξουσία. Το ακεί, το κεκτημένο, το κοινοτικό είναι αυτό το οποίο καλείται να διαχειρίζεται. Ενθυμίστε τι είχε γίνει στο παρελθόν με τη Μάργαρετ Θάτσερ και την ενιαία πράξη παρόλα αυτά υποχώρησε, δεν έθεσε βέτο, ο Μέιτζορ είχε υποσχεθεί πολλά κι όμως υπόκυψε και αυτός. Είδαμε τι γίνεται, είδαμε τι γίνεται με την μετανάστευση. Πράγματι νομιμοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αν οι πρωθυπουργοί δεν είχαν βάλει τις υπογραφές τους δεν θα βρισκόμασταν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Ο κύριος Βιτορίνο αναφέρθηκε στο ένας επίτροπος μία ψήφος στην Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι οι 18 της Ευρωζώνης θα υπερισχύουν πάντα των 10 εκτός και σχετικά με τις ομάδες αυτών που θα ασχολούνται με θέματα εξωτερικά, ομάδες επιτρόπων που θα ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα. Για φανταστείτε όλοι αυτοί να είναι από την Ευρωζώνη σε μια ομάδα, τότε θα συμπαρασύρουν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι θα κληθούμε να υπηρετήσουμε την Ευρωζώνη και τι αντισταθμίσεις θα υπάρξουν, δεν το βλέπω. Εδώ να μιλήσω σαν παράδειγμα πάλι με την κοινή αγροτική πολιτική που έχει ξεκινήσει η συζήτηση εδώ και δύο χρόνια. Τέσσερις εκθέσεις, 8.500 τροπολογίες, η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου ζητήθηκε και από το Κοινοβούλιο ε, φυσικά ο Ιρλανδός Επίτροπος ή μάλλον ο Υπουργός Γεωργίας της ε, Ιρλανδίας σε ένα δείπνο χόρεψε στο τραπέζι για να προκαλέσει τη συμφωνία των συμπολιτών του. Παρ' όλα αυτά πίστεψαν ότι συμφώνησαν και μετά φτάσανε στις λέξεις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συμφωνία, αλλά παρόλα αυτά έχει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αλλάξει απολύτως αυτό στο οποίο είχαμε συμφωνία. Καταλαβαίνω βέβαια ότι όταν υπάρχουν χιλιάδες τροπολογίες δημιουργούνται κάποιες αμφιβολίες νομικές για τη διατύπωση του κειμένου. Αλλά έβαλαν άσχετα πράγματα μέσα όπως ε, τα επιδοτούμενα πρόβατα έπρεπε να είναι θηλυκά. Εμείς δεν το είχαμε πει ποτέ αυτό. Το θέμα είναι και ότι εμείς δεν μπορούμε να τροπολογήσουμε τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και δεν μπορούμε και να τις απορρίψουμε και έχουμε προθεσμίες για την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα και δεν ξέρουμε πόσες ακόμα εξουσιοδότηση πράξης θα υποδεχθούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς θα αντιδράσουμε σαν Ευρωβουλευτές ε, λόγω των χρονικών ορίων. Αν πούμε ότι τις απορρίπτουμε θα χρειαστεί να ξανάρθουν πριν από τις εκλογές και τότε θα επιτρέψουμε σε μια μεταρρυθμιστική διαδικασία να προχωρήσει στην οποία δεν είχαμε ποτέ συμφωνήσει. Ε, και θα προτιμήσουν κάποιοι βέβαια να αποτύχει η διαδικασία παρά να πούν την αλήθεια ε, στους ε, εκλογείς τους και αυτοί είναι που προωθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουμε συνεχώς έκτακτες συναντήσεις της τελευταίας στιγμής και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και με τον Δεκάστρο και τον Επίτροπο Τσίολος και τίποτα δεν βγαίνει ακόμα. Είμαστε σε πλήρη αβεβαιότητα. Νιώθουμε ότι μας, έχουν, μας την έχουν στήσει γενικά και δεν πρόκειται να βρεθεί μια σωστή λύση για όλους. Καλώς φτάνουμε στο τέλος του χρόνου σε αυτό το κομμάτι της συνεδρίασής μας πριν από την απάντηση του κυρίου Βιτορίνου έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Μπρόνς. Ακούσαμε ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε στα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών για το διορισμό του Προέδρου. Μα αρχικά ε, ε, είχαμε πει ότι θα ορίζονται εναλλακτικοί υποψήφοι για την Προεδρία και στη συνέχεια θα ψήφιζαν οι ψηφοφόροι για μία λίστα, ε, ίσω με του ΕΛΚ, α πούμε, μια ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα και επί τη βάση αυτή τη λίστα θα διορίζονταν υποψήφοι για την Προεδρία. Όμω το κοινό δεν έχει καν ακούσει για τι λίστε των ευρωπαϊκών πολιτικών πολιτικό Δεν οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει η Επιτροπή. Αφήστε, μην μιλήσουμε καν για τους ε, Ευρωπαίους Επιτρόπους. Δεν ξέρουν ε, ε, τι σημαίνει η Προεδρία και δεν ξέρουν ούτε, ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, ούτε καν γνωρίζουν τίποτα για αυτές τις λίστες. Τώρα, το αν θα επηρεαστεί η ψηφοφορία από τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών, ότι θα βασιστούμε στην απόφαση του εκλογικού σώματος ε, που αγνοεί ε, το εκλογικό σώμα. Δεν έχει κανένα νόημα. Ε, μιλήσατε για τους ευρωπαϊκούς δήμους εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπάρχουν συναρθρεί που θα μπορούσαν να παραλληλιστούν με τους Δήμους. Τέλος πάντων δεν υπάρχουν τέτοιοι ευρωπαϊκοί Δήμοι, αλλά και να υπήρχαν ε, δεν συνδέονται με αυτές τις λίστες ε, των ευρωπαϊκών κομμάτων. Ε, στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να συσχετιστούν με την λίστα της, του Εθνικού Κόμματος. Ε, αυτό που έχω να καταγγείλω εγώ είναι η έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής και ενημέρωσης του λαού εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει κανένα άλλο το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στον ε, Επίτροπο, πρώην Επίτροπο, πώς να σας αποκαλέσω, Βιτορίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να ε, καταστρέψω το χρονοδιάγραμμά σας. Θα είμαι σύντομος. Θα διευκρινίσω ένα μόνο σημείο. η ιδέα του να ε, ε, οργανωθεί εσωτερικά Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της ιδέας των ομάδων επιτρόπων των κλάστερς σημαίνει ότι η συλλογικότητα δεν ε, λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Κοιτάξτε, όχι, ε, ε, δεν είναι ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από τις ομάδες των επιτρόπων, θα λαμβάνονται από το συνολικό σώμα των επιτρόπων. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή επίσημες αποφάσεις που θα λαμβάνονται από τις υπομάδες των επιτρόπων που θα εκπροσωπούν ενδεχομένω τι χώρε της Ευρωζώνης, παραδείγματο χάρη. Κύριε Άγνιο, ε, στην πράξη, ευχαριστώ την προσοχή σα στο ότι από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα 18 έχουν προσχωρήσει στο ενιαίο νόμισμα, δύο έχουν εξαίρεση, το δικό σας ε, κράτος μέλος και η Δανία, και άλλα 10 θα προσχωρήσουν αργά ή γρήγορα. Ε, στην Οπότε, στην πράξη, βάσει του κράτους δικαίου, η πλειοψηφία των κρατών μελών είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι στην Ευρωζώνη. Ε, ε, το εντελώς αντίθετο θέλω να εξασφαλίσω εγώ, το ότι η αποφάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εμβάθυνση τη οικονομική και πολιτικής ενοποίηση σε επίπεδο Ευρωζώνη, να φροντίσουμε να μην υπονομεύσουν το κοινό έδαφος της οικονομικής ολοκλήρωσης που κατ' εμέ είναι η ενιαία αγορά όπου εκπροσωπούνται και τα 28 κράτη-μέλη. Αν λοιπόν θέλετε να ε, διαστρεβλώσετε ε, και να ερμηνεύσετε εντελώ αντίθετη την δική μου άποψη σχετικά με τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ΟΝΕ, δεν ισχύει. Δηλαδή δεν πρόκειται να λαμβάνονται οι αποφάσει από υπομάδα επιτρόπων που εκπροσωπούν χώρε Ευρωζώνη. Όλοι οι επιτροπή θα εμπλέκονται διότι η ΟΝΕ είναι κοινή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παρότι ανάλογα με το στάδιο προόδου κάθε κράτους μέλους ε, υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί όροι για τη συμμετοχή αυτού στην Ευρωζώνη. Ε, η μνά μας η βασική είναι η λειτουργία της ενιαίας αγοράς να μην υπονομεύεται από περαιτέρω αποφάσεις για την εμβάνθυνση της ε, ΟΝΕ σε επίπεδο ευρωζώνης. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία για την ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του φίλου μου Πάλο Ραγγέλ. Ε, ευχαριστώ τον ε, πρόεδρο ε, Καζίνη και όλους όσους με άκουσαν σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ. Ο εισηγητή έχει ζητήσει το λόγο γρήγορα παρακαλώ, αλλά είστε εισηγητή βέβαια. Θα είμαι, είμαι σύντομο. Βεβαίω και θέλω να ευχαριστήσω για την συμβολή όλων των συντονιστών, πολύ σημαντική άλλωστε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Αντώνιο Βιτορίνο για την ανάπτυξη του θέματος και για τις απαντήσεις που έδωσε και να απαντήσω μόνο στον συνάδελφο Φόξ. <clears throat> Γιατί βρίσκω ότι στα λόγια του υπάρχει κάποια αντίφαση. Ως γνωρίζετε, υποστηρίζω την προσπάθειά σας για ενιαία έδρα. Αν όμως ισχυρίζεστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δημοκρατικό όργανο ή όχι ορθώς δημοκρατικό. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει. Εκείνο ορίζει την έδρα. Να αλλάξει τους ρόλους και να επιτρέψει το Κοινοβούλιο να επιλέξει έδρα. Ο λόγος για τον οποίο και εγώ αγωνίζομαι υπέρ μιας ενιαίας έδρας είναι διότι πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε δημοκρατικό όργανο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίζει το πεπρωμένο μας. Αν όμως πιστεύετε, όπως μας είπατε, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το πραγματικό δημοκρατικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει κανένας στόχος σε αυτή, τον αγώνα που κάνετε εσείς ο ίδιος να αλλάξετε τις έδρες και να τις κάνετε μία έδρα. Δεν έχει κανένα νόημα. Μόνο εάν πιστεύετε ότι είμαστε πραγματικοί εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών και ότι έχουμε την εντολή, τη σχετική εντολή τους, τότε θα πρέπει να είμαστε κυρίαρχοι να οργανώσουμε τις εργασίες μας όσο επιθυμούμε και να αποφασίσουμε ποια είναι η έδρα μας. Είπατε όμως εσείς σαφώς ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο εκπροσωπεί τους λαούς της Ευρώπης και όχι το Κοινοβούλιο. Ε, τότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ας αποφασίσει που θα πρέπει να συνερχόμεθα. Μια και αυτή είναι η κυριαρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα επομένως έχουν κάθε δικαίωμα να το πράξουν. Αυτά λοιπόν τα λόγια που λέτε και με τον τρόπο που σας τα ανέπτυξα αποτελούν αντίφαση και ήθελα να το πω. Αλλά κατά τα άλλα είμαι απόλυτα αλληλέγγυος μαζί σας στον αγώνα υπέρ μιας έδρας. Αλλά βέβαια για τους αντίθετους λόγους. Καλώς αυτό το πρώτο τμήμα λοιπόν της συνάντησής μας θα τελειώσει εδώ, το πρώτο πάνελ και θα ξεκινήσει το δεύτερο πάνελ στα πλαίσια του οποίου θα πάρουν το λόγο ο καθένας για 15 λεπτά ο διευθυντής ε, Νίμεν Κρίστενσεν, ο κύριος Μπόκμανς, Πάρξ, και μετά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Βιτορίνο για την παρουσία του και θα δώσω το λόγο στον Διευθυντή Κρίστενσεν για 15 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα αγαπητά μέλη που επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει κάποιες απαντήσεις στο πρόγραμμα της σημερινής συνάντησης. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η Γενική Γραμματέας, η κυρία Ντέιβις, δεν μπορούσε να είναι μεταξύ μας ε, σήμερα και θα μεταφέρω τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγώ. Το θέμα είναι αν καταρχάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τις νέες του αρμοδιότητες. Η εικόνα σήμερα δείχνει ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ εδώ και τέσσερα χρόνια η συνθήκη έχει επισκιαστεί δυστυχώς από την οικονομική κρίση. Το θέμα της διαχείρισης της οικονομικής κρίσης θα έλεγα ήταν ε, το πρωταρχικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα δεν ήταν ένα θέμα που αφορούσε 18 χώρες από τη μία και 10 από την άλλη. Η κρίση είναι τέτοια φύσεως που θα μπορούσε να διαλύσει το ευρώ και να υπονομεύσει την οικονομική σταθερότητα και όλων των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι Δανός και σε χώρες όπως και η Δανία θα είχαν χτυπηθεί άσχημα εάν πράγματι είχε διαλυθεί το σύστημα του ευρώ και αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια δηλαδή είναι ότι από τότε που συνετάχθη η συνθήκη στο Μάστριχτ η Ευρώπη, το ενιαίο νόμισμα, το ευρώ δηλαδή, θεωρήθηκαν σαν ένα βήμα προς την ολοκλήρωση. Είναι σήμερα σαφές ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα επιπλέον σημείο που, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά είναι ο κορμός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αυτό θα επηρεάσει το σύνολο της Ένωσης. Αυτό με οδηγεί σε κάποιες ε, σύντομες αντιδράσεις και σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο Άντζιου Νταφ. Το Συμβούλιο στα πλαίσια αυτού του περιβάλλοντος ίσως να έπαιξε έναν δυσανάλογα μεγάλο ρόλο να πω ότι εμείς συζητήσαμε το θέμα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και των νομισματικών πολιτικών, των 26 πρώτα και 28 μετά χωρών, σε τομείς που ανήκουν στις λεγόμενες εθνικές αρμοδιότητες. Δεν ήταν εύκολο λοιπόν να το ρυθμίσουμε αυτό και φάνηκε ότι ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση αντιστοίχων καταστάσεων στο μέλλον. Και αυτό το πετύχαμε χάρη και στον δραστήριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μέσω του εξαπλού και του διπλού πακέτου. Στα πλαίσια του εξαπλού πακέτου τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον νομικά την ε, ε, υποχρέωση να ελέγχει εκ των προτέρων τους εθνικούς προϋπολογισμούς πριν υιοθετηθούν, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία, η συνεκτικότητα τα πραγματικά έσοδα, τα πραγματικά έξοδα κτλ. Αυτός είναι ένας σημαντικός ρόλος, ένας ρόλος πολύ καθοριστικός θα έλεγα, που δείχνει ταυτόχρονα και την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στον τομέα του οικονομικού συντονισμού για την οικονομική σταθερότητα και την πρόβλεψη, πρόβλεψη των οικονομικών εξελίξεων. Βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο βέβαια στο οποίο τα κοινοβούλια των κρατών μελών παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι εθνικές δημοσιονομικές αρμοδιότητες δεν μπορούν να εξατμιστούν και γι' αυτό θα ήθελα όλους να σας ζητήσω να σκεφτείτε ε, για το πώς μπορεί κανείς να ενισχύσει τις σχέσεις ανάμεσα στα κοινοβούλια των κρατών μελών και τα ευρωπαϊκά όργανα και εσάς φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι τώρα υπήρχε μια αντιθετική, ε, αδικαιολόγητα αντιθετική σχέση ανάμεσα στα κοινοβούλια και σε εσά. Αλλά νομίζω ότι μέσω των συναντήσεων που κάνουμε τον τελευταίο καιρό ανάμεσα δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τμήματα επιτροπές των Κοινοβουλίων των κρατών μελών λειτουργούν καλά. Είναι σε εμβριακή ε, φάση στην παρούσα συγκυρία αλλά νομίζω θα βελτιώσουν τα πράγματα, ήδη έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μια επιπλέον προκαταρκτική παρατήρηση ε, είχαμε δύο κίτρινες κάρτες, ε, μηχανισμός επικουρικότητας. Οι δύο κάρτες αυτές. Η πρώτη ε, αναιρέθηκε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε την πρότασή της. Όχι λοιπόν αγνοήθηκε. Αυτό που συνέβη ήταν όταν εμείς σηκώσαμε την κίτρινη κάρτα, και είδαμε πώς θα εφαρμόζαμε την αρχή της επικουρικότητας, φάνηκε ότι ο τομέας τελικά απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο και υπήρχαν πάρα πολλές αρνητικές απόψεις και στο ίδιο το Κοινοβούλιο για την προτινόμενη μεταρρύθμιση. Συνεπώς λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρήθηκε από τις υπηρεσίε μας χαμένη πλέον και γι' αυτό και απεσύρθη. Δεν υπήρχε νόημα να επιμείνουμε μπορούμε να μπούμε σε μία σε βάθος ακαδημαϊκή συζήτηση για το αν έγινε σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας, αλλά δεν έχει σημασία γιατί απεσήρθη. Το δεύτερο θέμα αφορά τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα. Βλέπω εδώ διάφορα άλλα μέλη που είχαν συζητήσει το θέμα αυτό και την εποχή της ε, συνέλευσης για την Ευρώπη και υπήρχαν χώρες οι οποίες ε, είχαν αρνηθεί να εμπλακούν στην διαδικασία αυτή. Παρ' όλα αυτά είχε προβλεφθεί κάτι νομικά και οι 27 τότε χώρες, 28 τώρα, είχαν υπογράψει την ιδέα της δημιουργίας της θέσης ενός Ευρωπαίου εισαγγελέα. Και αυτό είχε προβλεφθεί και σε επίπεδο δημοσιονομικό. Ε, θα έλεγχε δηλαδή τις απάτες και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ο προϋπολογισμός δεν εφαρμόζεται σωστά κυρίως στα κράτη-μέλη και από τα κράτη-μέλη, αλλά παρόλα αυτά δεν θέλουμε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας να τα εξετάζει τα θέματα αυτά, θα το κάνουν οι χώρες μόνες τους. Αυτό δεν είναι σωστό. Απαιτείται ένας Ευρωπαίος Εισαγγελέας έτσι ώστε να υπάρχει μια ουσιαστική επίβλεψη της κατάστασης. Στην ουσία τώρα συγχαίρω τον κύριο Ράγκελ για τις ενδιαφέρουσες ιδέες της. Εμείς δεν ολοκληρώσαμε πλήρως ε, την επεξεργασία των θέσεών μας γύρω από τις προτάσεις Ράγκελ, αλλά είναι κάτι το οποίο λαμβάνουμε συνεχώς υπόψη μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό προκάλεσε πάρα πολλές ε, διαφοροποιήσεις. Το Κοινοβούλιο σφραγίζει ε, όχι μόνο τον προϋπολογισμό αλλά και τα θέματα αστυνομικής συνεργασίας, τα ποινικά θέματα, τα θέματα εξωτερικής ε, πολιτικής όπως επίσης και θέματα γεωργίας, αλληλείας κτλ. Πάρα πολλά θέματα πλέον και δεν θα αρνηθεί φυσικά να εφαρμόζει τις ε, αρμοδιότητες τις οποίες να ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει σε επίπεδο διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων όπως είδαμε στην περίπτωση του SWIFT. Έχουμε και το θέμα βέβαια της επόμενης, της εκλογής της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολιτικά. Θα μάθουμε το καλοκαίρι. Η ενίσχυση λοιπόν του Κοινοβουλίου από τη μία και η θεσμοποίηση του Συμβουλίου από την άλλη μετακίνησε την ισορροπία των εξουσιών στις Βρυξέλλες εις βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι, αυτό είναι λίγο πρωτόγονη σκέψη. Επειδή εσείς πήρατε πολύ, εμείς παίρνουμε υποχρεωτικά λίγο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ε, η πραγματικότητα αναγνωρίζει την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, την μονοπωλιακή πλέον ουσιαστικά δυνατότητα πρωτοβουλίας την οποία έχει και η αλλαγή του συστήματος των πυλώνων όπως επίσης και η αλλαγή των μεθόδων ψηφοφορίας και της στάθμισής του στο Συμβούλιο έχει καταστήσει τη λήψη των αποφάσεων ευκολότερη και διευκολύνει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μάλλον έχει ενισχύσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε ότι στους τριμερίους διαλόγους ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαν ειλικρινούς ενδιαμέσου βοηθά να βρεθούν λύσεις, κάνει προτάσεις και συνεισφέρει εν πάση περιπτώσει στην επίλυση των δυσκολιών. Όπως είπα λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όσοι πήρατε μέρος στην συνέλευση για την Ευρώπη, στόχος της συνθήκης ήταν να ενισχύσει όλα τα όργανα. Κανένας δεν είπε θέλουμε να εξασθενήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων ή τον ρόλο του Συμβουλίου. Ποτέ δεν ήταν αυτή η πρόταση της συνέλευσης. Η πρόταση ήταν να ενισχυθούν τα κομβικά όργανα στους τομείς αρμοδιότητας τους και να υπάρχει ισότιμη αντιπροσώπευση νομοθετική του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο και το βλέπουμε αυτό σήμερα να εφαρμόζεται. Συνεπώς λοιπόν το σύστημα το οποίο δημιουργήσαμε το σύστημα αυτό το ενωσιακό ή κοινοτικό πρέπει να είναι δημοκρατικό, πρέπει να είναι αποτελεσματικό και νομίζω ότι δεν ανησυχούν οι πολίτες ε, τους οποίους συνάντησα στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες για την ισορροπία των αρμοδιοτήτων. Αναφερθήκατε στις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Είναι αλήθεια ότι και η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Έχουμε τους ιδίους στόχους. Εσείς σαν Ευρωκοινοβουλευτική, εκπροσωπείτε τα πολιτικά σας κόμματα ε, στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όχι ανταγωνιστικά με το Συμβούλιο, αλλά το Συμβούλιο παρόλα αυτά αναζητεί τον κοινό παρανομαστή ανάμεσα σε 28 εθνικές θέσεις. Συνεπώς λοιπόν υπήρχε βάση για αυτήν τη νέα μορφή σχέσης ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και αυτό αντικατοπτρίζεται και στη νέα διοργανική συμφωνία την οποία διαπραγματευθήκαμε. Θα επιτρέψει τα όργανα να ξεκαθαρίσουν τους κανόνες σε διάφορους τομείς τους οποίους θα προϋπήρχαν συγκρούσεις. Ε, εδώ διαπιστώνω με χαρά ότι και τα κοινωνικά θέματα στο Συμβούλιο ε, δεν δημιουργήσαν πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση σαν παράδειγμα τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου στις ομάδες διαπραγμάτευσης των διεθνών συμβάσεων. Όταν λοιπόν αναφέρεται κανείς και στα θέματα του προγραμματισμού θα δείτε ότι η επταετής επόμενη περίοδος θέτει σε λειτουργία τις πρώτες φάσεις προγραμματισμού. Είχαμε ξεκινήσει τον προηγούμενο Ιούνιο μαζί σας, συναντηθήκαμε οι επίτροποι, συναντήθηκαν οι επίτροποι με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές Εμείς ε, προσπαθούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά. Ε, ε, σχεδιάζουμε την περίοδο που θα ακολουθήσει, περίοδο 12 μήνη, 16 μήνη, 18 μήνη, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε σαφώς την νομοθεσία. Αυτό αφήνει από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο μια χρονική περίοδο που προηγείται της κατάθεσης των τελικών προτάσεων. Η μοναδική ανησυχία εδώ είναι ίσως κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης η απουσία του Συμβουλίου Υπουργών και όχι μόνο στα πλαίσια της υιοθέτηση του 12 μήνου μάλλον προγράμματος. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει και μετά τους 12 μήνες και νομίζω ότι ο προγραμματισμός εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αλλά με ανησυχεί πάντα η αποσία του Συμβουλίου στη συγκεκριμένη περίπτωση και η μη εμπλοκή του. Είναι σαφές όμως για μας ότι ένα από τα νέα βασικά χαρακτηριστικά σε πολιτικό επίπεδο είναι η επίσημη ετήσια ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επηρεάζει και τα οργανικά θέματα αλλά και τις στρατηγικές επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο για την επόμενη περίοδο αλλά και ε, πιο μακροπρόθεσμα. Τώρα για τις πρωτοβουλίες επί τη βάση του άρθρου 225 Πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η συμφωνία πλαίσιο κωδικοποιεί το, το, το πώς θα γίνει αυτό. Στην ουσία όμως έχει υπάρξει κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έδωσε τις σωστές απαντήσεις. Δεν το κατανοούμε αυτό και δεν θα συμφωνήσουμε με αυτή την κριτική. Γιατί στην ουσία εμείς είχαμε μόνο 20 τέτοιες πρωτοβουλίες στις δύο τελευταίες περιόδους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ανταποκριθήκαμε στις μισές από αυτές, ε, σε έξι περιπτώσεις, όπως για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή για τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε άλλες περιπτώσεις εμείς αναγνωρίσαμε την εγκυρότητα των ετοιμάτων του Κοινοβουλίου αλλά επιλέξαμε διαφορετικά μέσα. Υπάρχει το θέμα της νομικής βάσης για τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης σαν παράδειγμα που υπάρχουν διαφωνίες αλλά αυτό είναι δευτερεύον, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι προσπαθούμε να απαντήσουμε μέσα σε τρίμηνη προθεσμία και να δώσουμε απαντήσεις ουσίας. Έχω προσωπική εμπειρία βέβαια από το ότι μερικές φορές οι βουλευτές οι οποίοι εμπλέκονται στην αρχική θεσμική εκκίνηση του 2025 δεν ενημερώνονται σωστά για την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι θέμα επικοινωνίας, ε, γιατί απαντούμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και όχι στους μεμονωμένους βουλευτές. Πρέπει λοιπόν το δίκτυο επικοινωνίας να λειτουργήσει καλύτερα και οι βουλευτές ε, να γνωρίζουν συγκεκριμένα την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις δικές τους πρωτοβουλίες. Τελικά για την Επιτροπολογία Πρόεδρε. Και αυτό τέθηκε σαν θέμα. Η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιλογή των νομικών βάσεων δείχνουν ακριβώς την ανάγκη να διαβάσουμε σωστά τη συνθήκη και να μην αντιπαρατεθούμε πολιτικά και κομματικά. Πρέπει να σεβαστούμε τις, αρμοδιότητες της πολιτικές ημέν των δε. Θα πρέπει αυτές να είναι οι προθέσεις μας πίσω από το 2.90 και το 2.91. Είναι πολύ καλή η έκθεση Shire έτσι ώστε να υπάρξει κοινό και νομίζω ότι στο παρελθόν υπήρξαμε αδικαιολογήτως ε, αντιθετικοί. Νομίζω ότι βέβαια βρισκόμαστε σε άγνωστα εδάφη και νομίζω ότι οι προτάσεις ε, τις οποίες κάνουμε δεν ήταν και οι πιο κατάλληλες. Όσο προχωρά κανείς ε, στην γεωργία ή σε άλλους συγκεκριμένους τομείς, ξέρετε ότι οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν πάντα με τον ίδιο τρόπο τα οριζόντια αυτά θέματα όπως τα γνωρίζουμε εμείς. Και πολλές φορές βρίσκουμε κάποιες λύσεις πρόχειρες λίγο, οι οποίες θεωρούνται και δεν γνωρίζουμε αν μπορούν να εφαρμοστούν μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων ή όχι. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις, ελπίζω ότι θα βρούμε σε μια λύση και κατά τη διάρκεια της παρούσης κοινοβουλευτικής περίοδου ή στις αρχές της επομένης. Και δεν πρέπει να υπάρχει λόγος έτσι ώστε να ε, διαιωνιστεί το πρόβλημα. Τέλος θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τις συστάσεις τις σχετικές με τις ευρωπαϊκές εκλογές θα στηρίξουμε τα κράτη-μέλη και τα πολιτικά κόμματα έτσι ώστε οι πολίτες ε, να ενημερώνονται σωστά για τους δεσμούς ανάμεσα στα εθνικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά κόμματα. Έχει νόημα να συνδέσουμε, να δείξουμε ότι αυτά που συμβαίνουν σε κάθε χώρα ενδιαφέρουν με ένα αλλά δεν είναι τα ίδια τα οποία συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι οι πολιτικές ομάδες που σχηματίζονται επί τη βάση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους πολίτες που θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν κοινέ βάσεις, κοινά θεμέλια και αυτό οι πολίτες το κατανοούν αυτοί που συνάντησα. Ξέρουν τι είναι τα πολιτικά κόμματα, ξέρουν ποια είναι η στόχη τους κτλ. Και γι' αυτό κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις και στην έκθεση την οποία εσείς καταθέσατε. Καλωσορίζω και τις υποψηφιότητες των κομμάτων, ακούγοντας από τον κύριο Νταφ πήρα πληροφορίες. Από ό,τι φαίνεται τώρα υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αλλά αυτά θα ακούσουμε περισσότερα και θα ενημερωθούμε καλύτερα. Πάνω στις συζητήσεις για μας είναι τακτικής φύσεως στην παρούσα φάση. Μέχρι τώρα οι ευρωπαϊκές εκλογές ήταν πάρα πολύ εθνικές και σε επίπεδο κυβερνητικό και σε επίπεδο κομματικό. Πιστεύουμε όμως ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να αλλάξουν τα πράγματα και μέσω του υποψηφίου Προέδρου να αναπτύξουμε μια διάσταση διαμεθοριακή η οποία να αντικατοπτρίζει τις σημερινές ευρωπαϊκές προκλήσεις. Και αυτό θα επηρεάσει και το σχηματισμό των πολιτικών αυτών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το μέλλον των πολιτικών τους φυσικά, να υπάρξει δηλαδή μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή διάσταση. Τέλος, τρίτο τέλος, θέλω να σας δώσω την εγγύηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να αναζητεί λύσεις με την κοινοτική μέθοδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία αυτή. Δεν είμαστε πάντα ικανοί βέβαια να επιβάλλουμε τις προτάσεις μας αλλά οι παλαιότεροι γνωρίζουν ότι μερικές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη κάνουν μια παράκαμψη και δεν πηγαίνουν στο άγνωστο αλλά περνούν σε κάποιες μορφές συνεργασίας διακυβερνητικές. Κατά καιρού τα είδαμε αυτά και γνωρίζουμε ότι μετά από 5-10 χρόνια λειτουργίας τους οι μορφές αυτές είναι λιγότερο αποτελεσματικές, λιγότερο χρήσιμες και επιστρέφουμε στην κοινοτική μέθοδο γιατί δουλεύουν καλύτερα. Δεν δουλεύουν τέλεια, αλλά δουλεύουν καλύτερα από τις εναλλακτικέ λύσεις. Συνεπώς λοιπόν προσπαθούμε να λύσουμε τα θέματα με την κοινοτική μέθοδο, παρόλα αυτά κάθε τόσο απαιτούνται κάποιες οριμότερες εξελίξεις και εκτός αυτής. Ε, ε, ε, το κύριε Διευθυντή, για το ίδιο θέμα Θα ακούσουμε τώρα και τους άλλους ομιλητές για την σχέση δημοκρατίας και κρίσης στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσον η κρίση έφυξε τη δημοκρατία. Ο κύριος Μπλόκμανς έχει το λόγο. Uh, uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πρώτα που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω ορισμένες από τις απόψεις του ΣΕΠΣ, του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών εδώ στις Βρυξέλλες, όπου μια ομάδα υψηλού επίπεδου εκπονεί εκθέσεις για τα θεσμικά μέσα στα πλαίσια της παρούσας συνθήκης. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται και ευρωβουλευτές και πρώην επίτροποι και άλλοι εμπειρογνώμονες. Στην παρουσίασή μου δεν απηχώ απαραίτητα τις απόψεις που περιλαμβάνονται στις εν λόγω εκθέσεις και οι οποίες θα δημοσιευτούν τον επόμενο μήνα. Έχω και μια παρουσίαση PowerPoint για ορισμένα από τα πιο εμπειρικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει. Η εφαρμογή των συνθήκ, της συνθήκης της Ένωσης μέσα από τη διαχείριση της κρίσης άνοιξε τα παλιά ερωτήματα και νέες προκλήσεις για την δημοκρατική νομιμοποίηση του συστήματος της Ένωσης. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που μου ζητήσατε είναι να αναφερθώ στα πιο κέρια θέματα και ως πανεπιστημιακός θα παραμείνω σε αυτήν την γραμμή και θα μιλήσω για πολιτική λογοδοσία και θεσμική ισορροπία εξετάζοντας τις εξουσίες που μοιράζονται τα όργανα μεταξύ τους σε τρεις βασικές φάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Έναρξη, εφαρμογή και, έναρξη ψήφιση και εφαρμογή. Για να αρχίσουμε από την αρχή, από την έναρξη. Τρία σχόλια εδώ. Η θεσμοποίηση και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και διαχείριση της κρίσης έχουν οδηγήσει στην διαμόρφωση των ε, εξουσιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γίνονται τώρα πλέον πολύ περισσότερες συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τρεις τον χρόνο, για μεγάλα θέματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τρεις έχει φτάσει σε 7 φορές τώρα να συνέρχεται το χρόνο και όλο και περισσότερο υπησέρχεται σε θέματα της καθημερινής άσκησης πολιτικής. Οι συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στρέφονται κυρίως από το, γύρω από τομείς πολιτικής που έχουν αναπτυχθεί εν μέρη ή και πλήρως εκτός της κοινοτικής μεθόδου. Διότι είναι ευκολότερο από άποψη εκχώρησης πολιτικής ιεραρχίας των χωρών. Οι συνθήκες του Μάστριχτ, Άμστερνταμ και της Λισαβόνας έδωσαν κεντρικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο συντονισμό της οικονομικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, της εξωτερικής πολιτικής, δικαιοσύνης και εσωτερικών, απασχόλησης κλπ. Παρ' όλα αυτά, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αφιερώνουν σημαντικό χρόνο και στις συζητήσεις άλλων θεμάτων υπό την κοινοτική μέθοδο, ιδίως περιβάλλον και ενέργεια. Και βέβαια και θα τα συζητήσουν αυτά και τον Μάρτιο. Η τάση αυτή έχει επηρεάσει και το ρόλο της Κομισιόν στην φάση της έναρξης της πρωτοβουλίας. Δεύτερο, η Κομισιόν εξακολουθεί να φέρει βασική ευθύνη για την πρωτοβουλία, ιδίω στα πλαίσια της κοινοτικής μεθόδου. Επόμενη διαφάνεια. Παρόλες τις προσπάθειες της Κομισιόν να μειώσει τον όγκο των νομοθετικών προτάσεων, ανακοινώσεων και άλλων εγγράφων, ο αριθμός τους εξακολουθεί να παραμένει υψηλό. Περίπου 700 πρωτοβουλίες ανά έτος εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 25% είναι νομοθετικές προτάσεις. Αυτά τα λέει η ίδια η ιστοσελίδα της Κομισιόν. Μέχρι τώρα η Επιτροπή Μπαρόσο έχει εγκρίνει 556 νομοθετικές προτάσεις και πάνω από 1100 άλλου ε, χαρακτήρα. Το γράφημα δείχνει την εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Η υπερβολική αυτή νομοθετική ε, πρωτοβουλία μειώνει την ποιότητα κάνοντας έτσι την εφαρμογή των προτάσεων δυσκολότερη. Η οργάνωση και λειτουργία του Συλλογικού Σώματος των, των ε, ε, Επιτρόπων, του λεγόμενου κολεγίου, όπως είπε και ο κ. Βιτορίνο προηγουμένως, μειώνει, α, μάλλον αυτά και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος μαζί είναι κρίσιμα στοιχεία για τον έλεγχο του ε, κριτηρίου της πρωτοβουλίας. Θα μιλήσω κυρίως εδώ βέβαια για τον έλεγχο της επικουρικότητας η συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας από πλευράς ε, θεσμών αλλά και ο έλεγχος από τις εθνικές βουλές είναι ουσιώδη για να αποφεύγεται η περιττή νομοθετική εργασία. Μετά από τέσσερα χρόνια χρήσης έχουν εντοπιστεί κάποια ελλείμματα και στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης των, ε, των Εθνικών Βουλών. Το 2012 η Κομισιόν έλαβε 83 συνολικά αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις που θεμελιώνουν την ε, παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας για 34 ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες, σημαντικότερο αριθμό δηλαδή από το 2010 και 2011. 24 κοινοβουλευτικά σώματα έστειλαν τουλάχιστον μία τέτοια αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Το 2012 τουλάχιστον οι μισές υποβλήθηκαν από τέσσερις βουλές, Σουηδική, Γαλλική και Ολλανδικές, πρώτη και δεύτερη βουλή, κάτω και ανωβουλή. Αυτά για το 2012, έτσι. Λέχθηκε ότι με την εξαίρεση της προτάσεως Μόντι 2, όλες οι υπόλοιπες νομοθετικές προτάσεις έλαβαν λιγότερες από πέντε γνωμοδοτήσεις και στη Μόντι 2 12 βουλές διαπίστωσαν παραβίαση της, αρχικής, της ε, αρχής επικουρικότητας, επομένως ε, έδειξαν κίτρινη κάρτα και οδηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τον Ιανουάριο του 2013 την πρόταση. Επίσης κίτρινη κάρτα εγέρθηκε πρόσφατα όταν 14 νομοθετικά σώματα προέβησαν σε ένσταση για το ε, αξιώμα του Ευρωπαίος Αγγελέος. Όμως η ε, Κομισιόν συνεχίζει με την ενισχυμένη συνεργασία στη βάση του άρθρου 96 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όμως αυτό δεν διορθώνει βέβαια την... αυτό που ισχυρίζονται δηλαδή οι βουλές ότι έχει υπάρξει παραβίαση της αρχής επικουρικότητας. Άρα δεν είναι σαφή τα πράγματα από την περιορισμένη εμπειρία που έχουμε ακόμα με τη χρήση του συστήματος Δηλαδή υποβάλλονται μεν αιτιολογημένε γνωμοδοτήσει από τις βουλές, παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνεχίσει την νομοθετική τη διαδικασία, απαντά στις βουλέ, αλλά δεν είναι σίγουρο αν λαμβάνει υπόψη τι απόψει του. Ορισμένε εθνικέ βουλέ μάλιστα παραπονούνται ότι οι επιστολέ απαντήσεω που λαμβάνουν από την Επιτροπή είναι πολύ γενικόλογε και δεν αναφέρονται στι συγκεκριμένε ενστάσει του. Τα ελλείμματα αυτά μπορούν να αποθαρρύνουν την επικοδομητική συνεργασία πολλών εθνικών βουλευτών και δεν υπάρχει και κοινή προσέγγιση στην αρχή της επικουρικότητας στο εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές βουλές συνήθως προβαίνουν σε ευρύτερη ερμηνεία της αρχής της επικουρικότητας και πολλά νομοθετικά σώματα θεωρούν ότι η αναλογικότητα είναι και εντάσσεται και μέσα στον έλεγχο της επικουρικότητας και οι περισσότερες αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις τελικά δεν ορίζουν πραγματικά την παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας και συνήθως έχουν πολιτικά κίνητρα. Ορισμένα, ορισμένες παρατηρήσεις τώρα για τις άλλες φάσεις, την διαπραγμάτευση και την έγκριση. Και πρώτα τον ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στην νομοθετική διαδικασία. Η χρήση της διαδικασίας συναπόφασης που δίνει κέριο ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την, ενίσχυ, για την ε, συμμετοχή του μεγαλώνει μέσα στα πλαίσια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας που καλύπτει 83 τομείς πολιτικής και μειώνει πλέον την χρήση ειδικών νομοθετικών διαδικασιών. Το επόμενο γράφημα της ε, παρουσίασης δείχνει ότι η συνήθις νομοθετική διαδικασία υπερτερεί των άλλων διαδικασιών. Μόνο στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας ε, λειτουργεί το Συμβούλιο χωρίς την συναπόφαση του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε ορισμένα άλλα θέματα σε ζητήματα εσωτερικών και δικαιοσύνης. Οι ειδικές διαδικασίες που απαιτούν σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μέτρα κατά των διακρίσεων και άλλα σχετικά, το ε, αξίωμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέως και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βέβαια, από την άλλη μεριά υπάρχει η διαδικασία του προπολογισμού, όπου όπου το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ε, προχωρήσει σε συνδιαλλαγή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον αυτό το τελευταίο δεν συμφωνήσει με τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ως αποτέλεσμα, ο ενισχυμένος ρόλος του Κοινοβουλίου ε, μέσα στην διαδικασία έχει προκαλέσει και νέες προκλήσεις διαθεσμικές. Τώρα, η επόμενη διαφάνεια πάλι δείχνει ότι για να αντιμετωπιστεί ο φόρτος εργασίας και να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις, η λήψη αποφάσεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στη, συνήθεια, στη τακτική δηλαδή νομοθετική διαδικασία επικεντρώνεται γύρω από ανεπίσημους τριμερείς διαλόγους και μάλιστα έχουν αυξηθεί οι συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση όπου απαιτείται μοναχά απλή πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει τις προτάσεις του, το Συμβούλιο μάλλον, να εγκρίνει τις προτάσεις του Κοινοβουλίου με ειδική πλειοψηφία. Γι' αυτό και υπάρχει τάση να καταλήγουν σε πρώτη ανάγνωση. Ενώ σε δεύτερη ανάγνωση απαιτείται απλή πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αλλά και άλλη πλειοψηφία στο ε, Συμβούλιο πολλές προεδρίες του Συμβουλίου ενισχύουν ενεργά τις συμφωνίες πρώτης αναγνώσεως. Όμως περισσότερο έλεγχο διαθέτει το Συμβούλιο αν προχωρήσει σε δεύτερη ανάγνωση. Διότι η κοινή θέση είναι η πρόταση για περαιτέρω διαπραγμάτευση και απαιτείται βέβαια και η δική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνδιαλλαγή και η τρίτη ανάγνωση ενδεχομένω εφόσον καταλήξει αδιέξοδο η δεύτερη ανάγνωση έχει πλέον σχεδόν εγκαταλειφθεί εκτός από ειδικέ διαδικασίες του προϋπολογισμού. Οι διαπραγματεύσεις σε τριμερή διάλογο διευκολύνουν και κάνουν πιο αποτελεσματική την μέθοδο ως ό,τι αφορά την σωστή χρήση του χρόνου, αλλά υπάρχουν και παρασκηνιακές συζητήσεις οι οποίες μειώνουν την πολιτική αξιοπιστία λόγω του ότι είναι μικρός ο αριθμός και είναι πολύ συχνά και γραφειοκράτες αυτοί που συμμετέχουν στους σχετικούς διαλόγους. Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τώρα. Η συνθήκη της Λισαβόνας διατάσσει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί νομοθετικές εξουσίες. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ορισμένες περιπτώσεις έχει υπερβεί τα όρια της συνθήκης της Λισαβόνας, για παράδειγμα για την οικονομική διαχείριση ή διακυβέρνηση. Επίσης, έγκριση συμφωνιών χωρίς λήψη υπόψη του θεσμικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και αν λάβει κανείς υπόψη ότι και το Ευρωπαϊκό Συμβολίο συμμετέχει και στην, Ευρωπα... και στην ε, νομοθετική διαδικασία ως συντονιστής ή επιβάλλοντας μια ε, επιλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του είδους είτε δέχεστε είτε την αποσύρουμε. Δεν είναι λοιπόν διαφανής η διαδικασία και περιθωριοποιεί εν μέρη και τους υπουργούς. Η αυξημένη δε δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι διότι γίνεται προσπάθεια να υπερβούν τις ε, τα εθνικά εσκαμμένα και είναι πολύ απίθανον κατά τη γνώμη μου η επιρροή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μειωθεί και πάλι στα προηγούμενα επίπεδα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν έχει κατακτήσει νέα εδάφη και, και μένει σε αυτά. Όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή λοιπόν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε, αλλά δεν έχει ενισχυθεί από την άλλη μεριά και το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, αποδίδει λόγο αντί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διευρυμένη διάσκεψη πρόεδρων πολιτικών ομάδων. Είναι πολύ περιορισμένες οι πληροφορίες που δίνονται εκ των προτέρων. Λαμβάνει μια έκθεση το Κοινοβούλιο μετά. Και ο πρόεδρος της Eurogroup δεν λογοδοτεί ούτε καν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ο έλεγχος των εθνικών κοινοβουλίων έχει αποδυναμωθεί σημαντικά σε πολλές χώρες μέλη. Εφαρμογή, φάση εφαρμογής. Υπό το φως νέων μέτρων που υιοθετούνται για την αντιμετώπιση νέων κρίσεων και ιδίως των νέων δημοσιονομικών και μακροοικονομικών κανόνων Ακόμα για την διάλυση τραπεζών θα τα αφήσω για τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Όσον αφορά την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων σε νέο σύστημα εποπτείας των τραπεζών, ακόμα αυτή είναι ανεπαρκής. Παρόλο που στις διαπραγματεύσεις του εξαπλού και του διπλού πακέτου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτυχε να περιλάβει τον λεγόμενο οικονομικό διάλογο και η αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσκαλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και του Συμβουλίου και όπου αυτό είναι ορθό και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο του Eurogroup να εμφανιστούν ενώπιον της για να συζητήσουν ορισμένα θέματα και αποφάσεις που έχουν ληφθεί στη διάρκεια του έτους, του έτους στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας. Τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει τις νομοδοτήσεις που δίνει και από τις κυβερνήσεις των χώρων της Ευρωζώνης και η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως και η Εθνική Βουλή μπορεί να προσκαλέσει εκπροσώπους της Κομισιόν ή των δύο τραπεζών που συμμετέχουν στον οικονομικό διάλογο και ταυτόχρονα διεξάγονται και διαπραγματεύσεις για την ώρα για ατομικές ρυθμίσεις συμβατικής μορφής με τα θεσμικά όργανα για μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχολήσεως. Στα πλαίσια αυτά, οι ατομικέ αυτές ρυθμίσει εγκρίνονται από το Συμβούλιο στη βάση προτάσεως της Κομισιόν. Το ΔΕ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην εκπόνησή τους, αν και θα έχει ρόλο στην εφαρμογή τους, εφόσον αναλαμβάνει και την εφαρμογή του τον έλεγχο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Συμπεραίνοντας τώρα, η φυστάμενη θεσμική ισορροπία έχει επηρεαστεί από την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην λήψη των αποφάσεων. Η δημοκρατική, ωστόσο, νομιμοποίηση και στο επίπεδο της Ένωσης και στο διεθνές επίπεδο δεν έχουν αυξηθεί αλλά μειώνονται και πρέπει να αυξηθούν στο μέλλον. Αυτό πιστεύω. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ. Κλείσαμε το πρώτο αυτό κομμάτι και δίνουμε το λόγο στον καθηγητή Πάρξ. Πριν από την τελική σύνθεση, την οποία θα κάνει ο επόμενος καθηγητής. Έχει το λόγο ο καθηγητής κ. Πάρξ. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα αρχικά. Ε, ε, ε, σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί ε, ε, θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεύτερον, αγνοήστε την ε, προφορά μου, γιατί μιλώ εξ ονόματος οργανώσεων της, μάλλον της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ με τις ερωτήσεις και να προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε απάντηση ε, στην ερώτηση σχετικά με το αν τα δημοκρατικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύονται μόνο και μόνο από ε, το ότι διαρωτούνται κάποιοι αν υπάρχει πλήρης άσκηση των αρμοδιοτήτων από πλευρά της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Κάποιες νέες εισαγωγικά χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπουν σε κάποιους ε, υπολογισμούς, στους οποίους θα σχολιάσω και μετά θα συνεχίσω. And the obvious one is interest representation. Ε, ισότιμη εκπροσώπηση, βασικό ζήτημα. Τα νέα κράτη-μέλη είναι ε, στην λάθος πλευρά ε, δύο βασικών χασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον πρώτον μικρές και μεγάλες χώρες και δεύτερον πλούσιες και λιγότερο πλούσιες χώρες. Αυτά είναι τα βασικά χάσματα που πλήττουν οποιοδήποτε ομοσπονδιακό σύστημα, οπότε πώς υπερεθνικά θεσμικά όργανα όπως η Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούν να καλύψουν αυτά τα χάσματα. Αυτό ενδιαφέρει τα κράτη-μέλη από πλευράς ισότιμης Σε Δεύτερη ερώτηση, η πορεία, ναι, είναι διαφορετική εστίαση. Υπάρχει το ερώτημα σε ποιο βαθμό τα δύο θεσμικά όργανα επιτρέπουν ε, στα νέα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να επηρεάσουν ε, τα πρότυπα που ε, εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν ε, τη διεύρυνση ήταν διαφορετικά τα, ε, τα πράγματα διότι δεν μετήχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θέλουμε όχι μόνο να συμμετέχουμε αλλά και να επηρεάζουμε τα τεκτενόμενα. Ε, τώρα, ε, κάτι που έχει αυξανόμενη σημασία είναι η διεθνή διάσταση. Δηλαδή, οι δημοκρατικέ αξίε Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποιο βαθμό προβάλλονται σε διεθνέ επίπεδο από αυτή την σκοπιά θα προσεγγίσω το ζήτημα. Δεν είναι ενοιολογική άσκηση, είναι ε, τρεις διαφορετικές οπτικές ε, γωνίες ε, που ταυτίζονται μάλλον με τις τρεις εκφάνσεις της νομιμοποίησης οποιοδήποτε δημοκρατικού συστήματος, δηλαδή υλοποίηση των συμφερόντων, δεύτερον οικονομική διαδικαστική νομιμοποίηση και τρίτον δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση και τέταρτον προώθηση των αξιών, δηλαδή αυτή η τέταρτη διεθνής διάσταση που σας έλεγα η προβολή των αξιών στο διεθνές επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε αυτά τα τέσσερα σημεία και κάθε φορά σε τρία υποσημεία. Ε, η ισότιμη εκπροσώπηση, αυτά τα ε, υπερεθνικά θεσμικά όργανα τελικά είναι πραγματικοί σύμμαχοι των κρατών μελών, όπως ε, νομίμως μπορούσαμε να προσδοκούμε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι βαθιά και ευρία η απογοήτευση, τουλάχιστον στι χώρε που εκπροσωπώ, σε σχέση με τι εξελίξει από τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα μέχρι σήμερα. Εκ πρώτη Θεωρήθηκε ότι πλήττει τα συμφέροντα των μικρών κρατών μελών η συνθήκη τη Λισαβόνα, αλλά με την κρίση και τι εξελίξει έχει ακόμη επιδεινωθεί η άποψη αυτή για την συνθήκη τη Λισαβόνα. Ε, θεωρείται ότι υπάρχει ένα κενό εξουσία σε σχέση με τον τρόπο ε, με τον οποίο τα θεσμικά όργανα ε, τρώνε το ένα τι αρμοδιότητε του άλλου, αν θέλετε αποδυναμώνεται τρόπον την έτσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενώ τελικά ε, βάσει των προτάσεων για τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, ενώ τελικά ενδυναμώνεται στην ε, ουσία και βλέπουμε ότι γίνονται στρατηγικές συζητήσεις ε, για την άμυνα το Δεκέμβρη, παραδείγματο χάρη οι επερχόμενες συζητήσεις για τη δικαιοσύνη και στις εσωτερικές υποθέσεις. Ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής συρρυκνώθηκε, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω πιέζει και συρρυκνώνει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αλλάξει και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τελικά όμως ε, δημιουργείται ένα κενό εξουσίας ε, λόγω της σύγχυσης των αρμοδιοτήτων λόγω ε, της συνθήκης της Λισαβόνας για την ισότιμη εκπροσώπηση δεύτερο θέμα για τις χώρες που εκπροσωπώ ξαναλέω το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωζώνη καλείται να καλύψει αυτό το κενό εξουσίας με υποπεριστάσεις διαφοροποιημένης ε, ολοκλήρωσης ε, και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μεγάλη δυσαρέσκεια σε σχέση με την αντίδραση από πλευρά του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιστάθηκε ίσως ε, στην ιδέα του ξεχωριστού προϋπολογισμού για την Ευρωζώνη, αλλά μόνο και μόνο ότι τέθη το ζήτημα και νομιμοποιείται ως εκ τούτου, αλλάζει την πορεία, αλλάζει την ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στην Ευρωζώνη και τις υπόλοιπες χώρες. Ε, υπάρχει λοιπόν απογοήτευση σε σχέση με, όπως είπατε και εσείς, το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν αναγνωρίζει την διαφοροποιημένη ολοκλήρωση και την πραγματικότητα ε, της ουσιαστικής συνεργασίας των κρατών μελών εκτός ορίων της συνθήκης. Υπάρχουν κάποιε βασικέ αξίε ε, με τι οποίε δεν συμμορφώνονται όλα τα κράτη-μέλη. Το δημοσιονομικό σύμφωνο δημιούργησε νέε νέες αρμοδιότητε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν νομίζω να κέρδισε από τι νέε αυτέ ρυθμίσει. Αυτό είναι το δεύτερο υπόσημείο. Ήθελα να σα πω ότι υπάρχει ε, απογοήτευση σε σχέση με την Ευρωζώνη που καλείται ξαναλέω να καλύψει αυτό το κενό εξουσία. Τρίτο σημείο, η πολιτικοποίηση ε, των σχέσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυξανόμενος ανταγωνισμός των δύο ε, που ε, αντισταθμίζεται με την ε, μάλλον ε, ε, πώς να πω, λιποβαρή σχέση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και, την, το Συμβούλιο. Τελικά το Κοινοβούλιο υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των νέων κρατών μελών γιατί υποφέραμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δηλαδή μπορεί να ήταν και προς μας που ανταγωνίζεται το Κοινοβούλιο το Συμβούλιο. με την σε Προεδρία ίσως να ε, ωφελεί αυτό σε σχέ... ως προς τις σχέσεις μας με το Συμβούλιο. Όμως ε, τελικά ε, το αποτέλεσμα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναλάβει να σπρώχνει τα βασικά ζητήματα και έτσι στερείται περιεχομένου το ε, Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων. Έχει δημιουργηθεί μια υπερκορεπέρ δηλαδή μέσα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, και επικρατεί ε, η ομάδα των χωρών της Ευρωζώνης. Σε σχέση τώρα με την εκπροσώπηση των συμφερόντων των χωρών και πώς αυτή επηρεάστηκε από τις διατάξεις συνθήκης Λισαβόνας και της κρίσης ε, είναι μάλλον αρνητική αξιολόγηση. Το δεύτερο ερώτημα οι πορείε, διαφορετικέ πορείε, ε, ο βαθμό των οποίων ε, οι χώρε τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τα νέα κράτη-μέλη μπορούν να επηρεάσουν τι υποκείμενε αξίε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξαναλέω, και εδώ είναι βαθιά η απογοήτευση των χωρών αυτών, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρείται ψυχικό σύμμαχο των νέων κρατών μελών σε σχέση με τροποποίηση των παλαιότερων αξιών, ε, μάλλον αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον αυτό πιστεύαν, όμω τα τελευταία χρόνια άλλαξαν τα πράγματα και πιστεύω ότι τελικά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει, συνάπτει ε, βραχύβιες, συνασπισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ερωτηματικά παραδείγματο χάρη για τον κανονισμό για τα προϊόντα καπνού, ε, ε, για τα ενεργειακά προϊόντα και τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που κάνει είναι ότι παραπαζαρεύει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βράχει πρόθεσμα. Για τον για την υπερβολική κοινοβουλευτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω ότι εξίσου υπάρχουν και ανησυχίες για την προεδρικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν ε, τελικά ε, ασκεί με ε, σωστό τρόπο τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναρωτιούνται τα νέα κράτη-μέλη. Η προεδρικοποίηση του συστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθεται όταν αναρωτιόνται για την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελικά φαντάζομαι ότι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι ότι αν δούμε και τι έγινε στην ε, περίπτωση του Επιτρόπου Ντάλι, ε, τελικά ο, Επίτρο... ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι υπόλογο σε σχέση με τα νέα αλλά και τα παλιά κράτη-μέλη. Για την ε, διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, ζητώ συγγνώμη αλλά έχουν αναφερθεί ήδη αυτά, τα βασικά μελλοντικά σημεία είναι η εφαρμογή των νέων συστημάτων, τουλάχιστον για τις δικές μας χώρες. Φυσικά θα παρακολουθήσουμε με προσοχή και ενδιαφέρον την πορεία της ε, Γερμανίας ε, το επόμενο εξάμηνο στην ε, Βαρσοβία τουλάχιστον επικρατεί η άποψη ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς τιμωρίας και κινήτρου για να εξευρωπαϊστούμε περισσότερο, αλλά θα πρέπει να δεσμεύονται όλοι ισότιμα από ένα αξιόπιστο σύστημα για την εφαρμογή, ε, επειδή είναι ένα είδος επιστροφής της απήχησης των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή μιλούσαμε και για την επιτροπολογία νωρίτερα, τα νέα κράτη-μέλη όχι μόνο μαθαίνουν ε, πώς λειτουργούν οι διαδικασίες, αλλά και διαπιστώνουν ότι στη δική μας χώρα δεν λειτουργεί αυτή η διαδικασία και επιστρέφει αυτό ως πληροφορία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την επιτροπολογία, λοιπόν, ε, πρέπει να αποφύγουμε την πολιτικοποίηση των εφαρμοστικών διαδικασιών και να μην αποτελέσουν οι νέοι κανόνες αντικείμενο διένεξη των θεσμικών όργανων, κυρίως σε μια εποχή όπου περιθωριοποιείται ο ρόλος τους. Σε σχέση λοιπόν με την αλλαγή των κανόνων και πώς αυτό ε, εφαρμόζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα ότι υπάρχουν σχετικά σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με τις νέες εξελίξεις. Το τρίτο ερώτημα τώρα. Η διεθνής διάσταση θα είμαι σύντομο. Θα είμαι σύντομος γιατί δεν θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό όπως τα δύο προηγούμενα σημεία, αλλά είδαμε σε σχέση με την Ουκρανία ότι είναι αυξανόμενη σημασία της διεθνούς αυτής διάστασης. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρόλα αυτά μπορεί να διαδραματίσει ένα ενδιαφέροντα ρόλο ε, στις διεθνείς σχέσεις ε, αν ε, επιλέξει τη σωστή οδό. Και πάλι τρία υποσημεία Υπάρχει απογοήτευση ε, σε σχέση με τις ε, ε, διενέξεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ως προς εξωτερικές υποθέσεις. Η Ουκρανία, νομίζω, η περίπτωση της Ουκρανίας δείχνει ότι δεν είμαστε σε θέση να έχουμε πλήρη πολιτικό συντονισμό για τις εξωτερικές υποθέσεις, για την αυξιακή βοήθεια, για την πολιτική γειτονία, για τη διεύρυνση, καλύπτονται όλα αυτά τα ζητήματα και επικρατεί η αίσθηση ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα μπορούσε πραγματικά να ενισχυθεί ούτω ώστε να μπορέσει να χαλιναγωγήσει τι πολιτικέ βλέψεις των κρατών μελών, κυρίως ως προ τι στρατηγικέ κατευθυντήριες γραμμές. Δεύτερο υποσημείο, ε, αναφέρθηκε ότι... Ε, ε, Ω προ τη συμπεριφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι υποψήφιε χώρε, παραδείγματο χάρη, Αναφέρθηκε λοιπόν ότι ε, ενδέχεται να ε, χρειάζεται να θεσπιστεί μια νέα θέση για τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αντιπρόεδρος υπηρεσίας εξωτερικής δράσης δηλαδή. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις πολιτικές ευαισθησίες των χωρών με τις οποίες συναλλασσόμαστε Δηλαδή, καλύτερα να ε, δούμε εκεί τα πέσα που έχουμε παρά να ε, τα επικεντρώνουμε στην, ε, στο, στην πλατεία Σούμαν. Ε, ενισχύοντας λοιπόν τον διαπραγματευτικό να της Ένωσης και προβάλλοντας τις δημοκρατικές αξίες της Ένωσης, βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καταλητική επιρροή σε εξωτερικό επίπεδο, τουλάχιστον σε επιχειρησιακό επίπεδο. Θα μπορούσαμε όμως να ενισχύσουμε το ρόλο μας ε, ε, σε άλλες δύο διαστάσεις των διεθνών διαπραγματεύσεων. Δηλαδή μπορούν Νομίζω ότι πλέον η υπηρεσία εξωτερικής δράσης αρχίζει να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εφάνει αυτό στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Εν κατακλείδη να κάνω και άλλες δύο παρατηρήσεις. Τελικά μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος ε, τι μας νοιάζει, ε, τι έχουν να πούνε για αυτά τα ζητήματα οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα νέα κράτη-μέλη. Θα απαντούσα το εξή. Οι χώρες ε, που μπήκαν με την τελευταία διεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά δεν έχουν προσχωρήσει με ολοκληρωμένο ε, τρόπο. Δηλαδή είναι εκτός κάποιων βασικών κανόνων και κάποιων κλειστών ε, ε, κύκλων ε, τώρα οι εντάσεις έχουν μετατοπιστεί ε, και διαπιστώνονται ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο και όχι ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή σε σχέση με αυτά που ήσχαν πριν από μία δεκαετία. Όταν μιλάμε όμως για πράγματα όπως η ελεύθερη κινητικότητα ε, ανακύπτουν και πάλι οι τάσεις ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή και στην επόμενη θητεία θα είναι ζητήματα που μας απασχολήσουν πάρα πολύ. Ε, πάντως ε, έχει αρχίσει να προκύπτει ένα θα το αποκαλούσα ανατολικό μπλοκ ε, σε σχέση ε, με τις ευαισθησίες ε, και τα προβλήματα που έχουν. Δεύτερον, υπήρξε μετατόπιση την τελευταία πενταετία σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πραγματεύονται όλα αυτά τα ζητήματα. Επικρίνουν πλέον την προηγούμενη άποψη που επικρατούσε ότι είναι φυσική του σύμμαχη το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχίζουν να επηρεασπίζουν τα δικά του συμφέροντα, τουλάχιστον στην Πολωνία, και αρχίζουν αρχίζουν να ποντάρουν περισσότερο στο διακυβερνητικό ε, πλαίσιο. Νομίζω ότι το ίδιο θα ίσχυε για το ζήτημα της τροποποίηση συνθήκης, παραδείγματο χάρη, ε, γιατί είναι ένας τρόπος, ε, θεωρούμε, να επαναπατριστούν κάποιες αρμοδιότητες από πλευρά κράτων μελών και η Πολωνία, παραδείγματο χάρη, θεωρεί ότι μπορεί να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο της διαφοροποιημένης προσέγγισης. Ένα τρίτο και θα κλείσω με αυτό. Ε, οι συζητήσεις ε, που γίνονται στην Πολωνία διαφέρουν ε, σε μεγάλο βαθμό από αυτά που συζητούνται εδώ. Δεν νομίζω το θέμα είναι η κοινοβουλευτικοποίηση ή η προεδρικοποίηση του συστήματος. Νομίζω ότι Μάλλον να συζητούμε την προεδρικοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την ε, διάχυση, το διασκορπισμό εξουσιών με την δημιουργία νέων ευρυδικών μορφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υιοθετώντα ε, διαφορετικές μορφές ευρωπαϊ... εναλλακτικές και πολλαπλές μορφές ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει εγγραφεί κάποιος... Βλέπω ότι ο συνάδελφος Νταφ θέλει το λόγο, θα μου έκανε εντύπωση αν δεν τον ήθελε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Νταφ, ευχαριστώ και αυτούς που πήραν το λόγο. Δεν σύμφωνο με όλα βέβαια, αλλά πολλά από αυτά που ακούστηκαν με βρίσκουν σύμφωνο και κάποιες από τις πρόπτικες που παρουσιάστηκαν. Τρία πράγματα. Πρώτον, Αυτό το οποίο μου λείπει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η έλλειψη στρατηγικής, ισχυρής στρατηγικής κατεύθυνσης. Κατά κάποιο τρόπο η εισβολή του Συμβουλίου σε αυτό το στρατηγικό επίπεδο διέσωσε νομίζω την Ένωση από την κρίση. Από την άλλη όμως δεν απέδωσε μια μακροπρόθεσμη συνεκτική κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο πετύχαμε αν θέλετε ήταν αυτός ο δικός χάρτης με την Τραπεζική Ένωση, την Δημοσιονομική Ένωση και την Πολιτική Ένωση. Αλλά και αυτός ο δικός χάρτης φαίνεται ότι έχει ήδη ξεχαστεί και δεν έχει αντικατασταθεί από κάτι άλλο από πλευράς του Συμβουλίου ή από πλευράς και της ίδιας της Επιτροπής Εδώ θα πρέπει να κάνω και αυτοκριτική βέβαια σαν, σαν κοινοβουλευτικός. Να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο εμείς λειτουργήσαμε και σκεφτήκαμε σε στρατηγικό επίπεδο ήταν ανεπαρκής. Και αυτό δείχνει αν θέλετε και την ποιότητα της ηγεσία των πολιτικών ομάδων και των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Συνεπώς θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να λειτουργεί σαν το πλέον πλήρες και αποτελεσματικό think tank στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν ιστορικά μόνο αυτός που προτείνει νόμους αλλά λειτουργήσε και σαν κίνητρο για τη διατύπωση κάποιων από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδέες. ιδιαίτερα στον τομέα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό το έκανε στο παρελθόν και ελπίζω στο μέλλον η Επιτροπή σύντομα να ξεκινήσει να το κάνει και πάλι. Τέλος, για τα κοινοβούλια. Ακούγεται περίεργο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι το κοινοβούλιο όμως δεν αντιμετωπίζει τις σχέσεις του με τα κοινοβούλια των κρατών με, με, αυστη, με σοβαρό τρόπο αλλά είναι σαφές ότι οι εμπειρίες που έχουμε από την Κοζάκ και τα λοιπά δείχνουν το επίπεδο της δυσκολίας. Τα κοινοβούλια των κρατών μελών δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερος ενήμερα των τελευταίων εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν ομόλογοι ιδίας αξίας. Και τα κόμματα των κρατών μελών, τα εθνικά κόμματα, ζηλεύουν θα έλεγα και αγνοούν ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Ένωση με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η δε αρχή της επικουρικότητας παρανοείται συστηματικά από όλους και δεν μας βοηθά και δεν είναι σίγουρα το πρίσμα μέσω του οποίου τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συνδέσουν τον εαυτό τους με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ευχαριστώ κύριε Νταφ. Ο κύριος Μπρόνς έχει ζητήσει το λόγο. Δεν υπάρχει και πολύς ανταγωνισμός. Ο καθηγητής Μπλόκμαν μας θύμισε, αν και δεν το χρειαζόμασταν, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τους προϋπολογισμούς τους στην Επιτροπή για έλεγχο. Αν και παραμένουν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών είναι υπεύθυνε στους εκλογείς τους για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, περισσότερο από κάθε άλλη ευθύνη που έχουν. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα πρέπει να θέσουμε σήμερα δεν είναι αν η κρίση έχει θέσει σε κίνδυνο τις δημοκρατικές, τα δημοκρατικά επιτεύγματα της Ένωσης, αλλά αν η απάντηση της κοινότητας στην κρίση έχει υπονομεύσει την δημοκρατία στα κράτη-μέλη. Καλώς. Έχουμε πάει πιο γρήγορα. Λόγω και της απουσίας του καθηγητή Εμμανουηλίδη και μπορούμε να ζητήσουμε από τους ε, προλαλήσαντες αν θέλουν να ξαναπάρουν το λόγο. Έχουμε 20 λεπτά ακόμα. Πριν κλείσουμε αυτή τη φάση της συζήτησης. Και θα ζητήσω μετά από τον καθηγητή Πέρνησε να κάνει την τελική σύνθεση. Θέλετε ξανά το λόγο. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα αυτή που μου δίνετε σχετικά με τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Εγώ συνεργάζομαι με τα Εθνικά Κοινοβούλια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συναντηθεί, Πρόεδρε, και στην Κοζάκα και στα άλλα πλαίσια. Έχει σημασία το θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Οι προτάσεις ε, δεν θα πρέπει να ε, κατατεθούν αν δεν έχει ελεγχθεί από τα κοινοβούλια η πλήρης εφαρμογή της αρχής επικουρικότητας. Νομίζω λοιπόν εδώ ότι ακόμα κανείς δεν έχει πει ότι δεν έχει ε, πάρει μια πλήρη αναλυτική απάντηση στην... Points We Απάντηση στην κίτρινη κάρτα για τον, ε, Ευρωπαίο Ισαγγελέα όπως ακριβώς ε, θα έπρεπε. Και αυτό γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι οι προτάσεις αυτές σέβονται πλήρως την αρχή της επικουρικότητας και μάλιστα προσωπικά μου είπαν ορισμένοι υπουργοί ότι οι απόψεις οι οποίες ακούστηκαν δεν ήταν ε, ένα θέμα απλά επικουρικότητας, αλλά ήταν μια αξιολόγηση της ιδέας για τη δημιουργία του, του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Να διαβάσετε την απάντηση, γιατί δείχνει ότι η κάρτα, η κίτρινη διαδικασία αυτή δουλεύει και το Κοινοβούλιο θα μπορέσει έτσι να συνεισφέρει και με την απάντηση του Συμβουλίου και να βρεθεί μια τελική απόφαση. Συνειδητοποιώ βέβαια ότι πολλές φορές οι εκπρόσωποι των κοινοβουλίων εδώ σήμερα στις Βρυξέλλες ε, μερικές φορές συγχέουν τα θέματα αυτά και αναφέρονται και στα θέματα της αιρεσιμότητας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και μπερδεύουν το θέμα με θέματα που δεν έχουν σχέση με την επικουρικότητα. Αλλά παρόλα αυτά οι απαντήσεις ε, ε, σίγουρα διαφοροποιούνται, σίγουρα υπάρχουν διαφωνίες, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το πιο σημαντικό θέμα είναι και σε σχέση με αυτά που είπε ο καθηγητής Πάρξ για αυτή τη νέα σχεδόν διαίρεση. Να είμαι ειλικρινής μαζί σας, εγώ δεν το βλέπω αυτό. Και δεν το βλέπω όχι γιατί δεν βλέπω το θέμα στο οποίο αναφέρατε, αλλά δεν έχουμε να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο. Ε, κάποιοι θεωρούν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να επηρεάσουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε στην Επιτροπή. Κοιτάξτε, ε, αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Είμαστε 28 χώρες. Ακόμα και οι μεγάλες χώρες αντιπροσωπεύουν η κάθε μία μόνη της μία μειοψηφία. Οι απόψεις λοιπόν οι οποίες ακούστηκαν από τα κράτη-μέλη είναι τόσο διαφορετικές που δεν υπάρχει μια κυρίαρχη άποψη. Άκουσα και τις απόψεις της Βαρσοβίας, Τι τις συγκρίνω με άλλες απόψεις εξίσου σημαντικές στην Πράγα, στην Πρατισλάβα ή αλλού. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε το ότι ζούμε σε ένα περίπλοκο οργανικό πλαίσιο. Όπως είπα είμαι δανός από μικρή χώρα. Οι μικρές χώρες προσπαθούν γιατί πάντα δεν επηρεάζουν όσο θα ήθελα να επηρεάσουν αλλά αυτή είναι η δημοκρατία. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε να κάνουμε με μία σύμπτωση, γιατί 7 από τις 10 νέες χώρες δεν ανήκουν ε, στην ε, Ευρωζώνη, ούτε στην αίθουσα αναμονής και προετοιμασίας για την Ευρωζώνη. Ελπίζω να κάνουν το βήμα αυτό να γίνουμε τον επόμενο χρόνο 19 και να υπάρξει και η Πολωνία στην Ευρωζώνη κάποια στιγμή. Είμαστε δεσμευμένοι λόγω της συνθήκης να μπείτε στο ευρώ όταν είσαστε έτοιμοι οικονομικά. Αν τα πράγματα πάνε καλά σημαίνει ότι τα προβλήματά σας θα εξαφανιστούν, ότι τα κράτη-μέλη θα ελέγξουν τις οικονομίες τους, ότι οι νέες χώρες θα μπουν στην Ευρωζώνη και θα συμμετέχουν στις διαδικασίες που θα λαμβάνονται για αυτούς. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συζητάτε και με τους Δανούς και με τους Βρετανούς, οι οποίοι εν τη σοφία τους αποφάσισαν να μην προχωρήσουν ε, στο ευρώ. Um, perhaps two words. firstly, because the question of national parliaments has come um, το θέμα των κοινοβουλίων έχει επανέλθει πολλαπλά. Η επανεμφάνιση των κοινοβουλίων στις συζητήσεις παρουσιάζει κάποιους κινδύνους και ο τρόπος με τον οποίο θέλουν να επιβάλλουν και να επηρεάσουν και να καλύψουν το δημοκρατικό έλλειμμα μπορεί να γίνει και μέσω της ενίσχυσης των εθνικών κοινοβουλίων που ελέγχουν τα θέματα της επικουρικότητας, της αποφάσεις της ευρωπαϊκές. Ίσως να υπάρχει μια έλλειψη επιθυμίας, αν θέλετε, να αντιμετωπιστούν τα, θέμα αυτά, τα θέματα αυτά σαν ευρωπαϊκά και τα βλέπουν περισσότερο σαν εσωτερικά. Ίσως αυτό να οφείλεται και σε έλλειψη συνεργασία σε επίπεδο ΚΟΖΑΚ. Ίσως ε, και λόγω της ε, παραβίασης της αρχής ή μάλλον της επιβολής της αρχής του πρίμους Ιντερπάρες από πλευράς του Bundestag να δημιουργούνται διαφορετικές συμπεριφορές. Θυμηθείτε τι έγινε στις συζητήσεις για τα bailouts όπου υπήρχαν δυνατότητες βέτο για βέτο από πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων που δεν φυσικά αναλήφθησαν ποτέ. Τίθεται λοιπόν το θέμα της εμπλοκής και του τρόπου εμπλοκής των Εθνικών Κοινοβουλίων στη συζήτηση. Ένα από τα θέματα τα οποία συζητήσαμε είναι το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη συζήτηση για τον διορισμό του Προέδρου της Επιτροπής και για τον συντονισμό των κομμάτων και τον ανταγωνισμό των κομμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. που θα καταλήξει στον διορισμό ενός υποψηφίου από τα κόμματα, κάτι το οποίο θα επηρεάσει θετικά, θα έλεγα, τη διακοινοβουλευτική συνεργασία και το λέω αυτό γιατί υπογραμμίζω ταυτόχρονα τη σημασία που έχουν τα κοινοβούλια των κρατών μελών στη συζήτηση. Για τη διαίρεση ανάμεσα στους παλιούς και στους νέους. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το έχουμε ίσως υπερβάλει παρουσιάζοντάς το. Στην ουσία το πρόβλημα είναι το αντίθετο από αυτό το οποίο παρουσιάστηκε. Όχι δηλαδή ότι τα νέα κράτη-μέλη φοβούνται ότι δεν έχουν αρκετή επιρροή, γιατί έτσι το βλέπει η Βαρσοβία σαν παράδειγμα, αλλά αυτοί που έχουν θα τους την πάρουν. Η βασική διαφορά είναι ανάμεσα στο βορρά και στο νότο και αυτό μας επιτρέπει εμάς στη Βαρσοβία να παίξουμε ένα επικοδομητικό ρόλο. Το θέμα είναι αν αυτό γίνεται αισθητό και το θέμα είναι ποιον δρόμο θα ακολουθήσουμε. Θα ακολουθήσουμε την διακυβερνητική οδό για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Α, ή θα ξεπεράσουμε το εθνικό κομμάτι και εμπόδιο και θα χρησιμοποιήσουμε την διεθνή συνεργασία και μέθοδο, την κοινοτική. Το θέμα δεν είναι η έλλειψη επιρροής λοιπόν, αλλά το πόσο σίγουρη και διαρκής θα είναι αυτή η επιρροή την οποία έχουμε. Τουλάχιστον έτσι το βλέπει η Βαρσοβία. Πολλές από τις χώρες αυτές λοιπόν έχουν την αίσθηση ότι αν και σε κάποια φάση θα μπουν στην Ευρωζώνη, ε, δεν θα ήθελαν να δημιουργούνται περισσότερα εμπόδια και το τέρμα να απομακρύνεται κάθε φορά που πλησιάζουμε, λόγω ακριβώς της περαιτέρω μείωσης ε, της σημασία μας η οποία πηγαίνει και το βάρος πηγαίνει προς τις μεγάλες χώρες της Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Ο Μπλόκμαν σε έχει να δώσει μια επιπλέον απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομη απάντηση στο πρώτο που ανέπτυξε ο κύριος Νταφ σχετικά με την πρόθεση ενός στρατηγικού σχεδιασμού. Σύμφωνοι, είναι πολύ σημαντικός και σημαντικό η έγκριση νέας νομοθεσίας να ανταποκρίνεται σε ξεκάθαρους στρατηγικούς στόχους, που βεβαίως θα έχουν θεσπιστεί εκ των προτέρων. Εν προκειμένου μια επικοδομητική πρόταση θα μπορούσε να είναι να προαχθεί, να προταχθεί μάλλον η νομοθετική διαδικασία ως σχεδιασμός, δηλαδή να προβλέπει η Κομισιόν ένα πενταετή σχεδιασμό που θα ελέγχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στρατηγικός λοιπόν νομοθετικός σχεδιασμός που θα, μπορεί, θα μπορέσει να συμβάλλει και στην αποτελεσματικότητα αλλά και στην ε, πολιτική νομιμοποίηση καθώς και στην διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Νομοθετικής Διαδικασίας επιτρέποντας άλλωστε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, έχει, ε, να υιοθετήσει μια πλέον μακροπρόθεσμη προσέγγιση και πιο ξεκάθαρους κατά προτεραιότητα στόχους. Με καλύτερη χρήση και των νομοθετικών εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας. Το ίδιο και ο ετήσιος διαθρωμένος διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προνομοθετικές αναθεωρήσεις που θα μπορούν να γίνονται έτος. Έχει ζητήσει το λόγο και ο συνάδελφος Σέπλιν. Yes, Thank you. Πράγματι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αν με επιτρέπετε να σκεφτώ λίγο έτσι φωναχτά πάνω σε αυτά που λέει ο κύριος Πάρξ. Ε, δεν ε, απευθύνομαι στην Κομισιόν βέβαια, δεν νομίζω να υπάρχουν κενά, ε, ε, απόλυτες, απόλυτα κενά ή απόλυτες διακρίσεις. Υπάρχει περισσότερο ε, μια ανάγκη να τοθεί διαφορετικά η έμφαση. Και μία από τις διαφορές που πρέπει να τονιστούν νομίζω και δύσκολο να βρεθεί αιτιώδη συνάφεια είναι το βάρος του κομμουνιστικού παρελθόντος. Όλες αυτές οι χώρες έχουν διαφορετική ιστορία από τις 15 αρχικές χώρες της Ένωσης που και αυτές βέβαια αποκλίνουν εννοείται. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι το δικό μας παρελθόν δεν ε, το ατενίζεται ως μέρος του ευρωπαϊκού παρελθόντος. Και γι' αυτό ακόμα μας λέτε νέες χώρες μέλη. Και αυτό κάτι συμβολίζει, κάτι δείχνει. Εφτά χρόνια είμαστε ακόμα οι νέοι. Πόσο καιρό θα είμαστε ακόμα νέοι, που να ξέρω ίσως για πάντα. Είναι ένα θέμα. Δεύτερο, και νομίζω τουλάχιστον αυτό οφείλεται εν μέρη ε, στην κρίση, αν δείτε την ιεραρχική σειρά των 27, γιατί εκεί τέτοιες στατιστικές είχα δει, για το ΑΕΠ ανακεφαλή. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο 2004 και στο 2012. Με άλλα λόγια, το 2004 η Σλοβενία, η Τσεχική Δημοκρατία ήταν μπροστά από την Ελλάδα και την Πορτογαλία Καμιά άλλη ανατολική νέα χώρα δεν έχει ξεπεράσει τις άλλες 15 παρά τα προβλήματα. Πάλι η Πολωνία και Ουγγαρία είναι πάνω μπροστά την Ελλάδα κτλ. Αυτό ε, είναι, αποτελεί μια ανησυχία και μια από τις δυσκολίες είναι η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων που έχει οδηγήσει σε μια φτώχεια στην εγχώρια συσσόρευση κεφαλαίου. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό, γιατί είναι και τέσσερις ελευθερίες και αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να εξετάσουμε την συζήτηση για τις ε, τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες, αν πραγματικά μπορούμε να μιλούμε για συζήτηση. Αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι μια μεταναστευτική κίνηση. Αν και βέβαια η ελληνική προεδρία αντέδρασε όταν είπα εγώ για ε, migration την προηγούμενη πέμπτη, η ελεύθερη διακίνηση τέλος πάντων, η ελεύθερη κίνηση αν αυτές λειτουργούν σωστά, διότι υπάρχει έλλειψη κεφαλαίου σε ορισμένες χώρες μέλη, ίσως υπάρχει από την άλλη μεριά η πλεονασματική προσφορά εργασίας και πάλι εκεί διστάζω να το χρησιμοποιήσω, αυτό όμως έχει σαφέστατες οικονομικές και κοινωνιολογικές επιπτώσεις. Το βρίσκω όμως απαράδεκτο ότι σε αυτές τις χώρες, τις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε δουλειές πολύ κατώτερες από αυτές που θα άρμοζαν στην εκπαίδευσή τους. γιατροί ή άλλοι πτυχιούχοι οι οποίοι δουλεύουν ως θηρορή ξενοδοχείων στο Λονδίνο. Το επόμενο που θέλω να πω είναι αυτή η συνεχιζόμενη συζήτηση. Μιλούμε για ανατολική γειτονία ή για σχέση με την ε, Νότια Ευρώπη. Εμείς θεωρούμε ότι η ανατολική γειτονία είναι πολύ σημαντική ιστορικά και κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε και μια διάσκεψη της Θεσσαλονίκης που να πει ότι αυτές οι έξι χώρες έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Με κάποιο τρόπο αυτές οι έξι χώρες που, σε οποίες αναφέρομαι, ανατολικά και νότια δηλαδή, πρέπει να έχουν μια ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν μπορούμε να τους καθυστερήσουμε για πάντα, διότι αν τους καθυστερήσουμε για πάντα κάποια στιγμή θα τις απορροφήσει η Ρωσία στη δική της σφαίρα επιρροής. Εν τέλει δε, δε όπως είπε και ο Δόκτωρ Πάρξ, ο πραγματικός πολιτικός φόβος ότι η Ευρωζώνη θα γίνει ο νέος πυρήνας της Ευρώπης από τον οποίο πάλι θα αποκλειστεί η κεντρική Ευρώπη. Και πάλι πρόκειται λοιπόν για μια ενδεχόμενη ιστορική εξέλιξη της ε, κεντρικής Ευρώπης. Και δεν είμαι βέβαιος ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης το έχουν αντιληφθεί αυτό. Θα ζητήσω λοιπόν από τον κοθήγητή Περνής, ο οποίος με πολύ μεγάλη υπομονή άκουσε όλες τις παρεμβάσεις, να μας πει τις βασικές του ιδέες, να κάνει τη σύνθεση της συζήτησης που προηγήθηκε και μετά θα κλείσει τη συζήτηση ο κύριος Βανζέλ. Έχετε όσο χρόνο θέλετε κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πρόεδρε. κυρίες και κύριοι, είναι... έχει περάσει η ώρα με προχωρημένη και έχουμε ακούσει πολλές και σημαντικές απόψεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να κάνω μια σύνοψη. Θα αντλήσω κάποια συμπεράσματα και θα σχολιάσω κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Η γενική μου παρατήρηση είναι ότι η συνολική συζήτηση, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι περί δημοκρατίας, περί του ρόλου ε, των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ιδιαίτερα, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις του Κοινοβουλίου σε σχέση με, την Επιτροπή, ε, με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Κάτι άλλο που δεν περίμενα να προκύψει στη συζήτηση είναι το θέμα της επικορικότητας. Η επικορικότητα είναι λένδετη με τη δημοκρατία μιλήσαμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Υπήρξαν θεμητές ανησυχίες ως προς την νομιμότητα των διαδικασιών και την παραβίαση επικουρικότητας και πιστεύω ότι και στην σημερινή συζήτηση και σε μελλοντικέ συζητήσεις θα πρέπει με πάσα σοβαρότητα και ε, να, εξηγήσουμε αλλά και να συζητήσουμε από πολιτικής πλευράς για ποιο λόγο χρειάζεται αυτή η διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταλαβαίνω πως για την περίπτωση του εισαγγελέα χρειάζεται, διότι αυτό προβλέπεται στη συνθήκη και συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να δοθεί συνέχεια λοιπόν σε αυτή την πρόταση. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις ίσως δεν ισχύει το ίδιο. Τι σημαίνει επικουρικότητα. Σε ποιο βαθμό η ύπαρξη ε, και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δικαιολογούνται. Είναι μεγάλη απόσταση και άρα η άμεση δημοκρατική συμμετοχή και επιρροή του λαού ε, στο ε, πολιτικό ε, γίγνεσθε είναι μικρότερη. Κυρίως όταν ε, ε, οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται σε πιο περιορισμένους κύκλους σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Λοιπόν, εάν ε, ανταυτού ληφθεί η απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς αυτή η δράση. Περί αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για την επικουρικότητα. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνει σε αυτό το απομακρυσμένο ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι. Για ποιο λόγο ε, δεν θα μπορούσε να ε, διευθετηθεί το ζήτημα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, Από την άλλη πλευρά, εάν εξηγήσουμε με ικανοποιητικό τρόπο, τότε δεν θα πρέπει να υπάρξουν λογικά καταγγελία σε εθνικό επίπεδο για την ε, εκχώρηση αρμοδιοτήτων, διότι δεν υπάρχει τέτοια εθνική αρμοδιότητα. Δηλαδή, εκχωρείται η αρμοδιότητα διότι δεν υπάρχουν τα μέσα σε εθνικό επίπεδο για να ε, υλοποιηθεί κάτι. Ε, μόνο έτσι ε, θα μας πάρουν στα σοβαρά. Δεν θα έπρεπε κάποιος βουλευτής να... Ε, ε απορρίπτει με την μεταβίβαση της αρμοδιότητας διότι δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι σε εθνικό επίπεδο. Μόνο εάν το αποδείξουμε αυτό μπορούμε ε, να νομι... μπορεί να νομιμοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι αρμοδιότητές της. Ε, ο κύριος Κάμερον όταν ναι, κατέθεσε τις προτάσεις του για την αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το ανέφερε και αυτό. Φυσικά, ε, εάν δεν είναι κάτι αναγκαίο, δεν θα πρέπει να υπάρχει. Κάποια αρμοδιότητα, αν δεν είναι αναγκαία, δεν πρέπει να υπάρχει. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω διαπιστώσει να συμβαίνει αυτό. Αλλά η συζήτηση σίγουρα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ε, σε μια τέτοια συζήτηση για τη δημοκρατία άλλο βασικό ζήτημα είναι πώς ε, οι επιθυμίες, η βούληση των πολιτών ε, θα μεταφραστούν σε δράσεις του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια πώς, σε ένα δεύτερο στάδιο, Αυτά που πρεσβεύει το Κοινοβούλιο και πιστεύει ότι θα πρέπει να συναποτελέσουν το μελλοντικό πολιτικό πρόγραμμα θα μεταφραστούν σε πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή θα πρέπει να ε, ακούσει το Κοινοβούλιο, να γίνει μια συζήτηση γιατί πρόκειται για το τρίτο στάδιο πλέον όπου η Επιτροπή θα καταθέσει τις προτάσεις της ε, για αυτά τα ίδια ζητήματα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα συντάξει τις ε, ε, πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν τρία διαφορετικά στάδια μεταβίβασης πληροφοριών και τα τρία θα πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Ε, σε αυτά θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας από τους πολίτες, ε, στο Κοινοβούλιο, από το Κοινοβούλιο στην Επιτροπή, από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μεταβιβάζονται οι πληροφορίες και θα πρέπει να προσέξουμε αυτά τα τρία διαφορετικά στάδια. Στην περίπτωση της ΟΝΕ αληθεύει πως για τις οικονομικές ε, πολιτικές το ε, πεδίο αρμοδιοτήτων είναι μάλλον εθνικό. Ε, δεν έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνω μόνο δύο παρατηρήσεις για αυτό το ζήτημα. Οι κυβερνήσει των κρατών μελών ε, πρότειναν ε, μια συγκεκριμένη ε, λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυτά μας οδήγησαν εξάλλου και στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και στον Ενιαίο Μηχανισμό. Η λύση αυτή πια ήταν περισσότερη συνεργασία, ενισχυμένη συνεργασία. Αναρωτιέμαι εγώ, μπορεί αυτό να αποτελεί τη λύση δεδομένης και της τελευταίας εμπειρίας που είχαμε, ας το πω με απλό τρόπο. η λύση για να επιτύχουμε ε, την ειρήνη στην Ευρώπη ήταν η υπερεθνική δράση, όχι η περισσότερη συνεργασία. Ήταν ε, αυτό που αποκαλείτε εσείς ε, κοινοτική μέθοδο, τα νέα θεσμικά όργανα κτλ. Αυτή είναι η μέθοδος τώρα, για, το, η λύση που υιοθετήθηκε για το προηγούμενο πρόβλημα. Το νέο πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι ο τρόπος συνεργασίας για ε, τις ε, οικονομικές ε, και κοινωνικές πολιτικές. Δεν λειτουργεί πλέον αυτή η μέθοδος και ποια απάντηση μας δίνουν τα κράτη-μέλη ότι χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία για να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα λειτουργήσει αυτή η λύση. Έχουμε τη δέσμη των δύο, των έξι οδηγιών για την οικονομική διακυβέρνηση, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, με όλα αυτά επιτύχαμε κάτι που μόνο βραχυπρόθεσμα μπορεί να λειτουργήσει. Τι θα συμβεί όμως ε, εάν δεν συμμορφωθεί με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο ε, το κράτος μέλος, δεν συμμορφωθεί με τις ε, νέες διατάξεις, τις νέες ρυθμίσεις, τι θα συμβεί, τίποτα. Και πάλι επαφιέμεθα στην καλή βούληση των κρατών μελών και είδαμε από εμπειρία, γνωρίζουμε μάλλον ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτό έξω και το πρόβλημα με την κοινοτική μέθοδο. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Με ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόσουμε την κοινοτική μέθοδο, την τροποποίηση των συνθήκων, την αναθεώρηση των συνθήκων ε, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και την κοινοτική μέθοδο, ώστε να λειτουργήσει και στην περίπτωση του συντονισμού των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Κάτι χρειαζόμαστε. Έχουμε τη δέσμη των δύο και των έξι οδηγιών και τα υπόλοιπα μέτρα. και ε, ε, κατακρίνουν αυτό το θέμα διάφοροι όπως ο φιλόσοφος Χάμπερμας, αλλά Χρειαζόμαστε σε αυτό, σε αυτό το τομέα κάτι καινούριο ε, και η νομιμοποίηση δεν μπορεί να έρθει ούτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι για τον απλό λόγο ότι κανείς δεν φέρει απολύτω την ευθύνη και εξάλλου σε ποιον λογοδοτούν οι κυβερνήσει των κρατών μελών ε, για το ευρώ. Ελήφθαν οι αποφάσεις και βλέπουμε ότι λειτουργεί, ε, είναι, νομοποιούνται οι αποφάσεις, αλλά σε πιο πολιτικό, ε, σε πιο, με πιο κοινωνικό κόστος σε χώρες όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Χρειαζόμαστε εντατικοποίηση της ε, κοινοβουλευτικής ε, συμμετοχής. Ε, ο κοινωνικός διάλογος είναι ένα βήμα, αλλά δεν επαρκεί. Η πιο εντατική συνεργασία ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και τις Επιτροπή Προπολογισμών του Κοινοβουλίου ή των ε, Εθνικών Κοινοβουλευτικών Δημοσιονομικών Επιτροπών ε, μπορούν να νομιμοποιήσουν περισσότερο τις διαδικασίες όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο όπου ένα εκτελεστικό όργανο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρεμβαίνει στη δημοσιονομική διαδικασία των κρατών μελών. Εγώ είμαι Γερμανός και ξέρω πώς, ε, ποια είναι η άποψη του συνταγματικού μα δικαστηρίου για αυτού του είδου. Ε, τη ρύθμιση. Δηλαδή το προσχέδιο του προϋπολογισμού πρώτα διαβιβάζεται το εκτελεστικό όργανο των Βρυξελών πρωτού καν το δουν οι εθνικοί βουλευτές και μόνο μετά την ε, συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κατατίθεται το προσχέδιο στη Γερμανική Βουλή και καλείται επίσης να εφαρμόσει τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, προς το παρόν ε, γίνεται δεκτό αυτό, αλλά πολύ αμφιβάλλω αν μακροπρόθεσμα θα γίνει αποδεκτή ε, η λύση αυτή. Θα ήθελα να δείξω και άλλα τρία-τέσσερα υποσημεία. Η, η μη άμεση εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρώτα απ' όλα πιστεύω ε, είναι ένα σημείο που τονίζεται ε, στη που δεν τονίζετε μάλλον πολύ στην έκθεσή σας, καλύτερα θα ήταν να το ε, αφήσετε απ' έξω, διότι ε, μπορεί να διαφωνήσουν κάποιοι, αλλά νομίζω ότι θα αποδυναμώσει το ρόλο του Κοινοβουλίου και θα δημιουργήσει επίσης άλλες, άλλα προβλήματα που ίσως τώρα δεν διαβλέπετε σε εθνικό επίπεδο. και αυτό το έμαθα από την απόφαση για τη Λισαβόνα του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. όταν ξεδόθη η απόφαση συζητήθηκε το εξής. Εάν υποκαθιστάται η νομιμότητα του Εθνικού ε, Συντάγματος από την ε, νομιμοποίηση του νέου ευρωπαϊκού λαού ε, ε, και την έκφραση της επιθυμίας του μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ε, ένα κράτος ή ένα ομοσπονδιακό κράτος, τουλάχιστον ένα ενιαίο κράτος, το οποίο είναι απολύτως αδύνατο ε, βάσει του θεμελιώδους νόμου της Γερμανίας. Ε, μιλώντας λοιπόν για την νομοποίηση των πολιτικών αποφάσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ε, αντικαταστήσει ένας ε, ευρωπαϊκός λαός στο γερμανικό λαό και τη βούλησή του. Ναι, όταν μιλούμε ε, για την ισοτιμία ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Για την άμεση εκλογή λοιπόν του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χρειαζόταν ίση ψήφος και προσοχή. Δεν ενστερνίζομαι αυτό το συλλογισμό ούτε και ε, το συλλογισμό βάσει το οποίο αυτό αντίκειται στο Σύνταγμα της Γερμανίας. Όμως υπάρχει, είναι κάτι που οπωσδήποτε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ίσως σήμερα δεν είναι η σωστή στιγμή να συζητήσουμε ε, το ζήτημα της άμεσης εκλογής του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερο σημείο, η εκλογή του Πρόεδρου της Επιτροπής. Πιστεύω ότι υπάρχει ε, Δήμος, ε, δεν υπάρχει μάλλον Δήμος Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δημιουργηθεί κάτι άλλο ε, συγκρίσιμο ε, με την έννοια του Ευρωπαϊκού Δήμου, η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Για τον ευρωπαϊκό λαό πιστεύω λοιπόν πως οι πρωτοβουλίες ε, για τον ορισμό των βασικών υποψηφίων των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων για την Προεδρία της Επιτροπής αυτό θα μπορούσε να δώσει στους ψηφοφόρους, στους πολίτες, για πρώτη φορά στην ιστορία, την επιλογή, μια πραγματική, ουσιαστική επιλογή για ε, τους ανθρώπους και για τα πολιτικά προγράμματα, τις προγραμματικές δηλώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων και αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολίτες των κρατών μελών, λοιπόν, ε, με την ταυτότητα, τη νέα τους ταυτότητα των Ευρωπαίων πολιτών, θα έχουν πλέον ε, την επιλογή ανάμεσα σε πρόσωπα και πολιτικά προγράμματα. Πιστεύω πως Εάν είναι λογικά αυτά τα πολιτικά προγράμματα και αυτοί οι άνθρωποι υποψήφοι ε, αγωνιστούν για να κερδίσουν ε, στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό θα δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους πολίτες για να ε, νομιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνέχεια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη ψήφο τους ε, στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ε, λοιπόν, θα έπρεπε να ζητήσουμε από τις ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με σοβαρότητα. Είναι πολύ αργά τώρα για να αρχίσει μια τέτοια διαδικασία. Το ΕΛΚ πρέπει πρέπει να σπεύσει ε, για να ορίσει τουλάχιστον τον ε, υποψήφιο στην κορυφή της λίστας γιατί ξαναλέω μόνο έτσι θα κινητοποιηθούν οι πολίτες και θα ε, δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές ε, εκλογές. δεύτερον ή τρίτον, ε, συμφωνώ με τον πρώην Επίτροπο και συνάδελφο τον καθηγητή Βιτορίνο γιατί τα κλάστες, ε, τις ομάδες επιτροπών, κάποιο άλλο αντίστοιχο σύστημα ανά θέμα, δηλαδή μπορεί κάποιο πραγματικά να αναρωτηθεί τι κάνουν όλη την ημέρα κάποιοι επίτροποι, γιατί είναι επίτροποι, ποιο είναι το χαρτοφυλάκι όντως όμως ε, στο εστερικό μιας ομάδας, αν ε, δηλαδή ε, υποδιαιρεθεί η Επιτροπή ανά τομέα αρμοδιότητας και λειτουργήσουν αυτές οι ομάδες επιτρόπων, θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να μειωθεί ο αριθμός των επιτρόπων. Η Επίτροπη τι είναι, η διεπαφή ανάμεσα ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο και τον εθνικό πολιτικό βίο. Χρειαζόμαστε αυτή τη διεπαφή, χρειαζόμαστε τους επιτρόπους. Είναι ο δικός μας επίτροπος, δεν εκπροσωπεί τα γερμανικά συμφέροντα. Είναι ε, ανεξάρτητος ε, και αμερόληπτος και τουλάχιστον όμως μπορεί να εξηγήσει στην Επιτροπή, τι συμβαίνει στη Γερμανία και στη Γερμανία τι συμβαίνει στην Επιτροπή. Πολύ βασική λειτουργία για τους Επιτρόπους. Ω προ ε, την ε, εκλογή ε, των υπολείπων μελών της Επιτροπής. Τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών σε κάθε κράτος μέλος είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη και θα έλεγα μάλιστα ότι κάθε κόμμα σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει μία λίστα ε, για να ψηφίσουν όλοι για τους υποψηφίους για το ε, Κοινοβούλιο. Ο πρώτος υποψήφιος στην κορυφή της λίστας ε, του κόμματος που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα πρέπει ε, να ε, εξεταστεί ε, σοβαρά ως ο βασικός υποψήφιος για την θέση του Επιτρόπου αυτής της χώρας. Όχι απαραίτητα, όχι με αυτόματο τρόπο, αλλά τουλάχιστον να εξεταστεί σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο, διότι έτσι νομιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο και έχει μεγάλη υποστήριξη από την εκλογική του περιφέρεια. Τέλος, για αυτή την ιστορία της μεταβίβασης δεδομένων που σας έλεγα στα διάφορα επίπεδα, δεν είναι ε, μία νέα πρόταση, ε, αλλά θα ήθελα να καταθέσω και πάλι αυτή την ιδέα. Εάν ε, έχετε μία επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχει ε, συμφωνήσει ε, ως επιτοπλίστων για το πρόγραμμα εργασίας για την επόμενη πενταετία και ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής προσπαθήσει να εφαρμόσει αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχει συμφωνήσει το Κοινοβούλιο και στο, όμως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο βρεθεί αντιμέτωπος με ε, αντίθετη ε, αντίθετη πολιτική ισορροπία ε, σε σχέση ε, με την ισορροπία του Κοινοβουλίου, όπως η συγκατοίκηση στο γαλλικό πολιτικό σύστημα, τότε αναρωτιόμαστε με ποιο τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη πολιτική συνοχή ανάμεσα στους δύο διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς. Αντί να έχουμε έναν ε, δυσυπόστατο λοιπόν πρόεδρο της Επιτροπής που ταυτόχρονα θα λαμβάνει και την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μπορούμε να πούμε ότι ε, θα έχει το διπλό ρόλο της εκπροσώπησης Ένωσης προς τα έξω και ε, προς τα μέσα. και στη συνέχεια ε, θα μπορεί να απευθύνεται στο Κοινοβούλιο ε, και να ε, απαντάει σε ερωτήσεις με ποιο τρόπο, παραδείγματος χάρη, εφαρμόζεται αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι, ο ερετός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη αρμονία με τις κατευθυντήριες, ε, στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό δεν ε, το συζητήσατε, ήθελα κι εγώ όμως να ε, προτείνω να υποβάλω και αυτή την ιδέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Ευχαριστώ λοιπόν. Εγώ απλά κατήφθηνα τη συζήτηση, ε, δεν έθεσα ερωτήσεις, αλλά κάποιες ε, μου έρχονται στο μυαλό και θα μου επιτρέψετε να θέσω μία, αν μου το επιτρέψει ο Ραντζελ. Είπατε ότι δεν υπάρχει δήμος, δεν υπάρχει λαϊκή στήριξη. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να αλλάξει και σε ποιο βαθμό τα όργανα της Ένωσης μπορούν να δημιουργήσουν αυτόν τον Ευρωπαϊκό Δήμο. Κοιτάξτε, δεν πολύ κατάλαβα αυτό που είπατε γιατί δεν δουλεύει το ακουστικό και γι' αυτό θα ήθελα να μου επαναλάβετε την ερώτηση. Είναι άραγε δυνατόν να υπάρξει δημοκρατία χωρίς τον Δήμο, χωρίς τον λαό. μπορούμε να περάσουμε σε ένα αφηρημένο δημοκρατικό σύνολο. χωρίς πραγματικό πολιτικό έλεγχο από πλευράς του λαού. Υπάρχει ευθύνη των πολιτικών σε κάποιο κοινοβουλευτικό σώμα. Χωρίς ένα πραγματικό δήμο και χωρίς την ταύτιση του Δήμου με την δομή, και τις αρχές της δημοκρατίας, δεν θα το πετύχουμε. Αναφέρομαι περισσότερο uh, στον Χάλσταϊν. Το κράτος είναι ένα πρότυπο πολιτικής οργάνωσης και μάλιστα στην περίπτωσή μας έφερε με την ειρήνη αλλά απέτυχε εν πολλής να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Είναι άραγε η καλύτερη απάντηση στο πρόβλημα αυτό να δημιουργηθεί ένα κράτος ευρωπαϊκού τύπου. και να μπούμε στη λογική του υπερκράτους με ό,τι αυτό σημαίνει σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Ή μήπως η ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί ένα νέο πραγματικά σύνολο, ένα υπερκράτος, το οποίο όμως αποτελείται από μια κατασκευή πολυεπίπεδη με μοίρασμα των εξουσιών ανάλογα με τις ανάγκες σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. έτσι ώστε κάποια πράγματα να αποφασίζονται από τα θεσμικά όργανα σε κάθε επίπεδο και έτσι να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουμε. Μήπως αυτή η οικοδόμηση είναι αντίθετη με την ιδέα μιας ένωσης η οποία θέλει να έχει ένα ενιαίο λαό και μια ενιαία κυβέρνηση. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Η ένωση που έχουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη στο να την παρουσιάσουμε και να την εκθέσουμε. Και το να χρησιμοποιούμε τα παραδοσιακά σχήματα, τα κρατιστικά, δεν είναι τελικά φαίνεται ο σωστός τρόπος. Είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος ε, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης ή μήπως πρέπει να αναζητήσουμε διαφορετικές λύσεις. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει τη νέα λύση και ίσως θα πρέπει να δείξουμε καλύτερα τις αρετές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίπεδο της κατανομής και του μοιράσματο των αρμοδιοτήτων και όχι απλά του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων. Ένα σφαιρικό σύστημα πολυεπίπεδο. Καλώς. Περάσαμε σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος τα οποία θα ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο. Θα κλείσει τη συζήτηση ο συνάδελφος Ράντζελ. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους κύριους καθηγητές, τον κύριο Μπερνίτσο ε, τελευταίο, για τα ενδιαφέροντα λόγια που είπαν. Συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα της επικουρικότητας ως pilot concept όλου αυτού του μηχανισμού. Το πρόβλημα όμως είναι ότι θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα αν γνωρίζουμε ποια είναι η ουσία της επικουρικότητας. Αυτή η ε, επικουρικότητα είναι μια διαδικαστική έννοια. Αν όμως πείτε, καλά, συμφωνούμε ότι αυτή η αρμοδιότητα, η τάδε αρμοδιότητα δεν μπορεί να ασκηθεί παρά μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως μερικοί βγαίνουν και λένε όχι καλύτερα στο εθνικό, άλλοι λένε καλύτερα στο ευρωπαϊκό. Να λοιπόν τότε που προκύπτουν οι διαφορές. Είναι πολιτική αποφάση. Επίσης, συμφωνώ με την άποψή σας που λέτε αν δηλαδή εκλεγεί άμεσα ο ε, πρόεδρος της Κομισιόν, αυτό θα αποδυναμώσει το Κοινοβούλιο. Αυτό ίσως ορισμένοι δεν το έχουν αντιληφθεί. Αν δηλαδή γίνει ευθεία η εκλογή α, του πρόεδρου της Κομισιόν, πώς θα είναι υπόλογος στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και έχει γίνει και προδεκαετίας, δεκαπενταετίας μια Ολλανδική πρόταση ότι εκλέγεται ας πούμε ευθέως ο Πρωθυπουργό, αλλά μετά προσέρχεται και λογοδοτή στο Κοινοβούλιο. Ήταν όμως μια περίπλοκη πρόταση, περίπλοκη διαδικασία. Το πρόβλημα όπως εντοπίσατε εσείς είναι στην πραγματικότητα η σχέση με το Συμβούλιο. Αν όμως θέλετε ισχυρό πρόεδρο της Κομισιόν, χρειάζεται την εκλογή. Όμως τότε έχετε προεδρικό σύστημα με δύο κοινοβουλευτικά σώματα και το Συμβούλιο παραμένει ως απλό νομοθετικό σώμα που ταυτόχρονα, καλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βέβαια όχι μόνο αλλά και τα διάφορα συμβούλια υπουργών όπως ΕΚΟΦΗΝ, ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών κλπ. Αυτοί λοιπόν οι σχηματισμοί αυτές, οι μορφές του Συμβουλίου ταυτόχρονα νομοθετούν. Έχουν όμως και το ρόλο του indirizzo πολίτικο, δηλαδή είναι και πώς να πω, και επικεφαλής κράτους. Γι' αυτό έχουν το, δικαιώματα, το δικαίωμα να διορίζουν τον Πρωθυπουργό. Όπως σε ορισμένα συστήματα όπου υπάρχει Πρωθυπουργό που ε, απαιτείται να έχει και την εμπιστοσύνη του, της Βουλής και την εμπιστοσύνη του Προέδρου, του αρχηγού δηλαδή ε, κράτους. Να, για παράδειγμα στην Κύπρο πριν από το 1974 υπήρχε μια συλλογική προεδρία, ένα είδος προεδρίου δηλαδή. Και αυτό που έχουμε τώρα, ανάλογο σύστημα δηλαδή το πρόβλημα, βέβαια τώρα με το Συμβουλίο, δεν έχουν, είναι ότι δεν έχουν μόνο νομοθετικές αρμοδιότητες όπως μια ανοβουλή, αλλά έχουν ταυτόχρονα και αυτό το ρόλο του indirizzo πολιτικό δηλαδή της ε, ε πολιτικών κατευθύνσεων. Ενώ δηλαδή τα τεχνικά της εκτελεστικής ουσίας τα έχει η Κομισιόν, το ανώτερο πολιτικό επίπεδο βρίσκεται στο Συμβούλιο. Και ο Άντζο Ντάφ είπε ωραία αυτά όταν έδειξε ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Και για τους ελεύθερους μάλιστα αυτοί οι δύο τρόποι φαίνεται πως είναι ξεκάθαροι τώρα πια. Αυτό που θέλω να πω εγώ με λίγα λόγια είναι ότι δεν είναι τόσο το πρόβλημα να έχουμε δύο ε, νομοθετικά σώματα με διαφορετικές νοοτροπίες όπως έχετε και στη Γερμανία. Το λεγόμενο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, Bundesrat, που έχει λιωτικές πλειοψηφίες από την Bundestag και λιγότερη διαφάνεια βέβαια. Εδώ είναι αλλιώτικα πάλι τα πράγματα. Όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Γερουσία έχει περισσότερες εξουσίες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τώρα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, νομίζω πρέπει να δούμε τη σχέση με το Συμβούλιο. Εσείς προτείνετε την λύση να έχετε μια διτή προεδρία. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο αυτό. Δεν θα είναι μάλλον. Υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό και έτσι θα ολοκληρώσω με δύο παρατηρήσεις. Αφενός το επιχείρημα που λέει ότι προσέξτε το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας, το γερμανικό συνταγματικό όλα τα συνταγματικά δικαστήρια Κατά τη γνώμη μου, τα όσα προτείνουμε συμμορφούνται με το γερμανικό σύνταγμα. Και αν όχι, τότε να το αλλάξετε. Εύκολο είναι αυτό, έτσι. Να το αλλάξετε το γερμανικό σύνταγμα, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αυτό είναι το θέμα. Το απλό γεγονός ότι βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει τα συνταγματά μας χωρίς να αλλάξουν τα κείμενά τους. Πρόκειται για συνταγματική αναθεώρηση αλλά άτυπη. Verfassungsänderung στα γερμανικά. Γι' αυτό πρέπει να πω και αυτή η δεύτερη παρατηρήσή μου, συνεχίζει ο κύριος Ραμζέλ, ότι υπάρχει ένα σημαντικό θέμα. Δεν είμαστε τώρα σε αυτό το state model politics, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Καμιά φορά λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μιμηθεί τις ΗΠΑ και αυτό δεν είναι καλή λύση. Ναι, το πρόβλημα όμως είναι ότι οι χώρες μέλη δεν ισχύουν πλέον όπως ήταν. Δηλαδή το κράτος μετά από τις συμφωνίες Βεσταλίας έχει ήδη εξαφανιστεί. Όμως εμείς, εμείς όμως πιστεύουμε ότι συνεχίζεται. Αυτό που γίνεται λοιπόν κατά κάποιον τρόπο είναι είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα είδος πολιτικού μοντέλου, μοντέλου συγγνώμη, που πρέπει να το μιμηθούν οι χώρες μέλη. Είναι ακριβώς το αντίθετο δηλαδή. Πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς αυτό. Στο γερμανικό δόγμα περί κράτους, η παράδοση λέει λαός, κυριαρχία, έδαφος, επικράτεια. Όμως η επικράτεια δεν είναι πλέον τόσο σημαντική γιατί είναι αδύνατον να περιοριστούν όλες οι πολιτικές καθαρά σε μία επικράτεια. Άρα και η μορφή του κράτους έχει αλλάξει πλέον. Απαντώντας στον αγαπητό μας πρόεδρο κ. Κασίνη θα έλεγα ότι πιθανώς μετακινούμεθα σιγά σιγά προς ένα μοντέλο που να συνδέεται περισσότερο με το Μεσαίωνα όπου δεν υπήρχε ένα κέντρο που ήταν το κέντρο το μονοπόλιο του κράτους, της εξουσίας, της νομιμότητας και της και του φυσικού εξαναγκασμού. Αυτό όμως είναι αδύνατο τώρα πλέον. Μέσα στα όρια μας είναι αδύνατο να υπάρξει αυτού του είδους το κράτος. Δεν υπάρχει μονοπόλιο. Υπάρχει πολυαρχία. Βλέπε Εγγελ. Όπως είπε αυτός δηλαδή ο φιλόσοφος για, ο Έγελος για το Μεσαίωνα. Άρα λοιπόν μάλλον πρέπει να κινηθούμε αντίστροφα. Τα κράτη και το γερμανικό κράτος και το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο θα πρέπει να εμπνευστούν από την ευρωπαϊκή διαδικασία και ουχή το αντίθετο. Γιατί μέσα στις ίδιες τις χώρες μας, μέσα στα έθνη μας, μέσα στα κράτη μας, αλλάζουν οι δομές της εξουσίας. Και άρα λοιπόν πιστεύω η προσέγγιση θα πρέπει να είναι διαφορετική. Το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι το σύγχρονο και τα κράτη είναι απερχαιωμένα. Καταλαβαίνω ότι μάλλον πρέπει να ολοκληρώσω εδώ γιατί αλλιώ ε, με συνεπαίνουν τα λόγια μου και αρχίζω και οραματίζομαι. Καλώς. Ήταν πολύ πλούσιο το απόγευμα που προηγήθηκε. Τελειώνουμε εδώ. Σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλους. Όλοι πραγματικά μας είπατε πολύτιμα πράγματα. Θα συναντηθούμε αύριο στις 9.30. 9 με 9 και μισή οι συντονιστές και μετά θα συνεδριάσει η Επιτροπή. Ε, ευχαριστώ. Μικρός το δέμας αλλά